Okay. So good uh, afternoon. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ε, ξεκινήσουμε σιγά σιγά την συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Όπως ξέρετε, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση αυτής. Εγκρίνεται, ωραία. Δεν έχω ανακοινώσεις του Πρόεδρου και δεν έχω και τίποτα να πω για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Οπότε, περνάμε στα σημεία 4 και 5. Έχουμε εδώ τον κύριο Λούντβιχσον από του Σοσιαλδημοκράτε. τίτλοι... Ε, ο τίτλος είναι Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Κάρτας Υπηρεσιών που θεσμίζεται με τον οικείο κανονισμό. και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση που απευθύνεται στην Επιτροπή Όπως ξέρετε τον Ιανουάριο η Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων με στόχο να διευκολύνει την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Ένα από τα εν λόγω μέτρα είναι η εισαγωγή της ε, νέας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών, έτσι ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν να ολοκληρώνουν τις διοικητικές διατυπώσεις που απαιτούνται σε άλλα κράτη-μέλη. Η ΙΜΚΟ πρότεινε να απορριφθεί η, της, ε, η πρόταση της Κομισιόν και θα συζητήσουμε αυτή ακριβώς την πρόταση ο 7 λεπτά, οι τέσσερα λεπτά και αν έχουμε αρκετό χρόνο μπορούμε να κάνουμε και ένα γύρο της αιθούσης 2 ε, λεπτά οι παρόντες. Ο κύριος Λούντβιχσον έχει τον λόγο για 7 λεπτά να κάνει μια εισαγωγή στα σημεία 4 και 5. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι σήμερα αναγκαίο να προωθήσουμε την ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών στην Ευρώπη. Γι' αυτό χαιρετίζω τα μέτρα τα οποία συνεισφέρουν στην ε, ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών. Αλλά αυτό πρέπει να πηγαίνει χέρι με χέρι με την τήρηση υψηλών προδιαγραφών για εργαζόμενους, για καταναλωτές και βεβαίω αυτά να ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις. Η πρόταση για την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Κάρτας Υπηρεσιών μπορεί να διευκολύνει κατά την άποψη της Κομισιόν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών και παραδείγματο χάρη θα διευκολύνει την ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλη χώρα. Έχουμε λοιπόν αφενός έναν κανονισμό που αφορά την ουσία και από την άλλη έχουμε μια πρόταση οδηγίας ε, που καθορίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής. Η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει κάποια προστιθέμενη αξία σε αυτήν την πρόταση. Όπως όλοι γνωρίζετε εγώ δεν έχω πιστεί για το ότι ισχύουν αυτά. Επιπλέον συμφωνώ με αρκετά από τα σημεία κριτικής που έχουν ασκηθεί από εργοδότες, ε, συνδικάτα, αυτοί οι οποίοι δηλαδή θα πλήγουν περισσότερο από αυτήν την πρόταση. Λένε ότι η πρόταση αυτή δεν προσθέτει τίποτα. Παραδείγματο χάρη, γνωρίζω ότι ο τομέας των ασφαλιών έχει ασκήσει ρητή κριτική στις σχετικές προτάσεις της Κομισιόν και λέει πως βασίζονται σε λανθασμένες υποθέσεις και αν εφαρμοστούν δεν θα λειτουργήσουν και θα κοστίσουν πολλά χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Στον τομέα της οικοδομής υπάρχουν φόβοι ότι μια τέτοια ηλεκτρονική κάρτα θα προωθήσει τη μαύρη εργασία, την παράνομη εργασία, τα μπλοκάκια κτλ. Και έχουμε λοιπόν διάφορες αμφιβολίες και επιφυλάξεις, ε, τις οποίες πρέπει να λάβουμε σοβαρή, σοβαρά υπόψη. Και η πρόταση της Κομισιόν ε, έχει γύρει μια σειρά ζητήματα. Παραδείγματο χάρη λέει ότι εάν κάποιος υποβάλει μία αίτηση μπορεί να εκδοθεί μια τέτοια κάρτα ακόμα και αν το κράτος μέλος δεν έχει αρκετό χρόνο για να κάνει τους ελέγχους. Πρόκειται δηλαδή για μια υπονοούμενη έγκριση με την οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Επιπλέον ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα και το παράθυρο για καταχρήσεις εάν ε, το δεχόμαστε χωρίς επαρκής ελέγχους. Μετά έχουμε τον χρονικό περιορισμό που περιορίζει την ικανότητα των κρατών μελών να κάνουν σοβαρούς Κατόπιν η διάρκεια ισχύς της κάρτας αυτής επίσης είναι πρόβλημα. Γιατί ε, μπορεί τα στοιχεία τα οποία δηλώνονται να είναι ήδη πεπαλαιωμένα και πριν ε, εισαχθεί ένα νέο σύστημα θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως ε, μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι, οι επιδιωκόμενοι με έναν τρόπο. Και θεωρώ ότι εάν θέλουμε να εισαχθεί ένα νέο σύστημα, είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε διατυπώσεις σαφείς, απλές, για να πραγματοποιηθεί ο στόχος της νομοθεσίας. Η πρόταση αυτή όμως είναι υπερβολικά περίπλοκη και περιέχει διάφορες ασάφειες σε διάφορα θέματα κεντρικής σημασίας. Και το θέμα γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο από το ότι υπάρχουν διάφορα τεχνικά μέτρα έτσι ώστε δεν θα λειτουργήσει τελικά το πράγμα στην πράξη. Και τελικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του εάν υπάρχει όντως κάποια προστιθέμενη αξία σε αυτήν την πρόταση. Μιλάμε για εισαγωγή περίπλοκων διοικητικών δομών που δεν θα έχουν και κανένα νόημα στην πράξη και δεν θα υπάρχει και ζήτηση για αυτές. Δηλαδή υπάρχουν ήδη πολλά μέσα σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει ακριβώς να τα αναλύσουμε για να ξεκαθαρίσουμε το εάν μια ηλεκτρονική κάρτα προσφέρει τίποτα παραπάνω ή όχι. Και, επιτρέπετε μου, πρέπει να πω ότι εγώ θα ήθελα να προτείνω να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν. Από την άλλη, θα ήθελα να τονίσω ότι εγώ είμαι ανοιχτός σε μια επικοδομητική συζήτηση για να ακούσουμε το ότι ε, έχουν και οι σκιώδησίτες των άλλων ομάδων. ευχαριστούμε κύριε Λούτφιξον για την εισήγηση αυτή να δώσω το λόγο στον κύριο Ματούσο από το ΕΛΚ Σκιώδη. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις αμφιβολίες μας και τις δικές μου αμφιβολίες για αυτό που συζητούμε. Συμφωνώ απολύτως με τον ε, καθελή αρμόδιο εισηγητή. Το ερώτημα είναι πώς θα το χειριστούμε το θέμα αυτό στην ΕΚΟΝ. Έχω πολλές αμφιβολίες για την ε, αρμοδιότητά μας και πολλές ανησυχίες. Γι' αυτό ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεσης. Υπάρχουν αρκετά σημεία που θα μπορούσα να είμαι σύμφωνος, όπως η ανάγκη να καλλιεργήσουμε την προσφορά υπηρεσιών. Αυτό είναι πάντοτε θετικό, αλλά υπάρχουν πολλά σημεία που έχουν να κάνουν περισσότερο με την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Επαναλαμβάνω λοιπόν τι αμφιβολίε μου για τι δικέ μα αρμοδιότητε επί του θέματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κατανοητό. Για τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Λούνες. Ευχαριστώ. από πλευρά του συναδέλφου να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν μπορούσα να είναι στη σημερινή συνάντηση, αλλά μου έστειλε το σημείωμά του. Σε ό,τι αφορά την πρόταση και καθώ την μελετούμε, έχουμε ήδη κάποιε προκαταρκτικέ παρατηρήσει. Πρώτον, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ομάδα των συντηρητικών μεταρρυθμιστών έχει κάποιε σοβαρέ αμφιβολίε για τα ζητήματα που έχουν τονιστεί εδώ. Συγκεκριμένα την ε, ε, διάρκεια χωρί ημερομηνία λήξη των ηλεκτρονικών καρτών. Έπειτα το χρονοδιάγραμμα ώστε όλοι οι ετούντε για τι υπηρεσίε μέσω ηλεκτρονικών καρτών να ελέγχονται πραγματικά από τα κράτη-μέλη υποδοχή πρωτού, οι ηλεκτρονικέ κάρτε εκδοθούν επισήμω. Τρίτον, Πιστεύουμε ταυτόχρονα ότι η αιτιολόγηση της έκθεσης αυτής είναι ε, κάπως ε, μη ισορροπημένη και θα πρέπει να αναλύσουμε τις ευκαιρίες και τις θετικές πτυχές του κανονισμού που προτείνονται. Η διαρκής εξάλληψη φραγμών και προσφορά διασυνοριακών υπηρεσιών ε, σε όλα τα κατημέλη μπορεί να παράσχει προσθεθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή αγορά με σημαντική μείωση του κόστου λειτουργίας για τις εταιρείε και βελτιώνοντας τη δυνατότητα επιλογής στην προσφορά για τους καταναλωτές. Καταλαβαίνουμε ότι σε κάποια μέλη οι άνθρωποι αρχίζουν να, να αγχώνονται για το ΕΠ του, της χώρας τους, για τις ακριβές υπηρεσίε. Έχουν κάποια προστατευτική ε, στάση ως προς την δική τους εσωτερική αγορά. Το καταλαβαίνουμε αυτό το άγχος. Αλλά είναι ένας φόβος ότι θα υπάρξει μια εισβολή φτηνών υπηρεσιών από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Να σας θυμίσω όμως μια άλλες δύο πτυχές στη βασική πρόταση σε ό,τι αφορά αυτό το, αυτή τη διάσταση, υπάρχουν διατάξεις που δηλώνουν το κάθε μέλος αποδοχής μπορεί να φροντίσει να επιβάλλει εγχωρίως ε, διατάξεις και να αποφασίσει αν οι ετώντες μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες στην επικρατεία του. Άρα το κάτω μέλος μπορεί να αποφασίσει ένα περίπτωση και διατηρεί τη βασική αρμοδότητα. Μέσω τη ηλεκτρονική κάρτα επίση δεν θα επηρεαστούν οι ισχύουσες υποχρεώσει ε, των εργοδοτών, δεν θα επηρεαστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, οπότε από αυτό το φω η πρόταση του ηγετή απλώς να απορριφθεί η πρόταση τη επιτροπή συνολικά είναι κατά την άποψή μα πρόημη και αδικαιολόγητη. Η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών πιστεύει ότι τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν και μάλιστα εύστοχα εάν τροποποιηθεί το κείμενο σε συνεργασία με την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ε, για άλλη μια φορά, πιστεύουμε ότι μια τροποποιημένη πρόταση μπορεί να είναι ένα βήμα πρόοδου για να βελτιωθεί η αγορά υπηρεσιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι και πρόκληση και ευκαιρία. Να μην την πετάξουμε, να την εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία γιατί οι εταιρείε μπορεί να έχουν φόβους και άγχη αλλά οι, χώρες στα οι εταιρείε στα διάφορα κράτη μας κατοχώρες και ούτω καταξή θα ωφεληθούν πολύ. Οι καταναλωτές θα έχουν μεγαλύτερη επιλογή από περισσότερα μέρη και θα είναι ευγνώμονε εφόσον ε, εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα και για τα σχόλια του και του εισηγητούς σα. Νομίζω ότι κάποιο θέλει να μιλήσει εκ μέρου των φιλελευθέρων, όχι. Από την ΚΟΕ, όχι. Από του πράσινου κάτι βλέπω. Δεν είστε εισηγήτρια, αλλά μόλι μπορεί να μιλήσει. Ναι, όντω. Αντικαθιστώ την σκιώδη συγγητρία. Ευχαριστώ τον, ε, ε, σκιώδη, τον ε, αρμόδιο συγγητή και τους σκιώδης που, για τη συνεργασία τους. Η πρόταση για απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που μας βρίσκει μάλλον σύμφωνο και είμαστε στην ίδια γραμμή συλλογιστική. Στηρίζουμε προτάσεις που μπορούν να ευνοήσουν την καλλιέργεια τη ε, αγορά υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Όμω, τέτοιε προτάσει πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα κράτη-μέλη υποδοχή έχουν όλα τα μέσα στη διάθεσή του για να ελέγχουν την αγορά υπηρεσιών και να φροντίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών, ε, οι πάροχοι υπηρεσιών τηρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές τους. Πολλές φορές είναι διαφορετικά ε, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές ε, στις χώρες υποδοχής σε σχέση με τη χώρα του παρόχου και δεν θέλουμε να υποβαθμιστούν αυτά τα πρότυπα για τους καταναλωτές της Ευρώπης. Η πρόταση γύρει πολλές αμφιβολίες για μας, όπως η αρχή της Σιωπηρής Συμφωνίας. Δηλαδή, ο ετών μπορεί να ζητήσει ηλεκτρονική κάρτα στη χώρα προέλευσής του και να την ε, φέρει σε ισχύ αν το κράτος μέλος υποδοχής δεν αντιδράσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι ηλεκτρονικές κάρτες χορηγούνται για απεριόριστη διάρκεια από ό,τι φαίνεται. Οπότε έτσι δεν ρυθμίζεται το δικαίωμα να αποκτήσει κανεί ηλεκτρονική κάρτα. Ε, Ω προ τι η πρόταση θα επιτρέψει σε ασφαλιστές και άλλες εταιρείες διανομής να εναρμονίσουν το σύνολο των όρων κάλυψης των πελατών τους σε περίπτωση σύναψης ασφάλειας. Αυτό πρακτικά μπορεί να μην είναι εφικτό. Θα είναι δυνατό να έχουμε ένα τέτοιο ενιαίο έντυπο, μια ενιαία μορφή στα έντυπα των ασφαλιών. Θα έχει αυτό προστεθεμένη αξία κατά των φραγμών που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ενιαία αγορά. Για αυτού του λόγου, κατά πάσα πιθανότητα θα υποβάλουμε τροπολογία που καλεί του συναδέλφου να απορρίψουν αυτέ τι προτάσει όπω πρότεινε και ο ίδιο ο εισηγητή. Η Μισελ αναμένει τι συζητήσει με του υπόλοιπου και όλου για το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου και στην αίθουσα. Και στο ΚΑΤΣΤΙΑΙ έχω την κυρία Μπερέφ. Με ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την πρότασή του. Είναι βέβαιο ότι θα απαντήσει στον κύριο Μαρτουσέλο. Α, έφυγε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το απαντήσει, λοιπόν, αλλά θέλω να επαναλάβω τη σημασία που έχει για την Επιτροπή μας να υπάρξει μια τοποθέτηση από πλευρά μας για το θέμα, διότι στο επίπεδο της Επιτροπής, ε, ακόμη και χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς στο Συμβούλιο, είναι σαφές από τις συζητήσεις που έγιναν εκεί ότι θα έχει άμεσο αντίκτυπο πρόταση αυτή της ασφάλειας. Χωρίς να μιλήσω για την φορολογία που δεν αναφέρεται καν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την κοιτάξει επισταμένως η Επιτροπή μας. Ποια θα είναι τα φορολογικά συστήματα που θα ισχύουν για μια τέτοια ιονή απόσπαση. Διότι πίσω από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό υπόκειται. Ε, στον τομέα λοιπόν των ασφαλιών πρέπει να δούμε τα πράγματα με σαφήνεια και να τα πούμε με ειλικρίνεια. Ε, για να μπορεί να τα κατανοήσει ο καθένα. Από την πρώτη οδηγία για την εσωτερική αγορά στον τομέα των ασφαλιών έχουμε επιλέξει να εργαζόμαστε προ την εναρμόνιση. Και εδώ προτείνεται απλώ ένα σύστημα αμοιβέ αναγνώριση. Σε έναν τομέα όπου δεν υπάρχει κανένας προεδ... καμία πρόοδος ως προς την σύγκληση των συστημάτων και κανένα συνολικό σύστημα εποπτείας, επίβλεψης και το καθεξής. Από την άποψη λοιπόν ε, και την στενή, υπό την στενή έννοια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά την πρόταση του συγητή μας εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Η κυρία Σαντέρ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Εάν κάποιος άλλος βουλευτής θέλει το λόγο στο καθένα μου το πει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα απλώς να σας διαβιβάσω τις έντονες επικρίσεις ε, ε, που μου έθεσαν υπόψη οι συνάδελφοι για την πρόταση αυτή που έχει γεννήσει πολλές αμφιβολίες και κριτικές. Ακούσαμε κάποια από τα θέματα το πρόβλημα με τις ασφάλειες, το πρόβλημα με την ε, σιωπηρή ε, αποδοχή, συγκατάθεση, το πρόβλημα της απεριόριστης διάρκειας. Όλα αυτά είναι διάφορα προβλήματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Ε, τη βλέπουν με πάρα πολύ ε, κρίσιμη ματιά οι Ευρωπαίοι και συμφωνώ με τον εισηγητή στα σχόλια και τις Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανένα άλλο ε, το λόγο, να παρακαλέσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Λότβιξον, να συνοψίσει για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω δεν θα χρειαστώ τα δύο λεπτά, Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι ε, το θέμα αυτό είναι λεπτό και ευαίσθητο. Άκουσα τις ανησυχίες και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των υπολείπων. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που είπαν τη γνώμη τους. Προφανώ όλα αυτά τα ζητήματα χρειάζονται λίγο περισσότερη εμβάθυνση. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Ότι είναι αμφιλεγόμενη αυτή η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως σας είπα και προηγουμένως, συμφωνώ απολύτως να συζητήσουμε τις τροπολογίες που θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας με όλους τους κοιόδες ηγητές να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Το θέμα δεν είναι εύκολο να λυθεί. Ξέρω ότι γνωρίζει μεγάλες επικρίσεις. Τα ακούω κι εγώ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναδούμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρειάζεται επεξεργασία σε πολλά από τα σημεία της. Προσωπικά εγώ θα ζητούσα απόρριψη της πρότασης αυτής, αλλά είμαι στη διάθεσή σας πρόθυμος να το συζητήσω με τους σκιώδεις ηγητές για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να βελτιώσουμε. Και να δούμε και τις τροπολογίες που ενδεχομένως να έρθουν. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου θα κάνω ό,τι μπορώ για να διευκολύνω την κατάσταση. Για να μπορέσουν να συμφωνήσουν, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδες όλους και τα μέλη που συμμετείχαν στη συζήτηση. Σήμερα είναι 16 του μηνός, η προθεσμία ε, χειριστεί για τις 19 Οκτωβρίου, 9 Νοεμβρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσει στις 4 Δεκεμβρίου η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούτβιξον για την έκκληση που απευθύνεται. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα ένα διάλειμμα μέχρι το επόμενο σημείο που έχει προβλεφθεί για τις 4 παρατέταρτο. Λοιπόν, 15 λεπτά διάλειμμα. Ευχαριστώ. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κηρύσω και πάλι την έναρξη της συνεδρίασης μας, μάλλον επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση, σημείο 6, πλαίσιο για την ανάκαψη και εξηγένση κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Το σχέδιο έκθεσης κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο μετά από ακρόαση και συνεννόηση με τους σκιώδεις. 218 είναι οι τροπολογίε, Μεταξύ άλλων η έκθεση τονίζει τη διαφορά ε, μεταξύ σεναρίων πτώχευσης και μη πτώχευσης σε περίπτωση ε, επιταχυμένης μετάβασης από την ανάκαμψη στην εξυγίαση ε, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις opt-in διάσωσης των τραπεζών από τους φορολογουμένος και να υπάρχει μια προστασία από πελάτες και καθαριστές. Ε, το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει εγκρίνει τη γενική του θέση. Εμείς έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Απουσιάζει και η Σουίμπορν, η συγκήτρια η συνεισηγήτρια από του ECR. Θα δώσω το λόγο στον άλλο εισηγητή, στον κύριο Ιάκωβ Φον Βάιτσεκερ, για πέντε λεπτά παρακαλώ, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και η ΚΕΙΜΕΝ απουσιάζει, αλλά θα ήθελα εγώ να την ευχαριστήσω την απουσία της και ίσως κάποιος μπορεί να τα διαβεβάσει αυτά στην Gay Sweeper. Στην αρχή θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι είναι μάλλον απίθανη αυτή ε, η ε, συνεισήγηση ε, κάποιος από το ECR και κάποιος από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Παρ' όλα αυτά εργαστήκαμε σε πολύ ε, επικοδομητικό πνεύμα. Ήταν αγαστή η συνεργασία μας και προσπαθήσαμε να ε, συναντηθούμε και με τους κοιόδες ηγητές. Ξέρω ότι υπήρξε πίεση χρόνου. Τώρα περιμένουμε τις τροπολογίες τους. Τώρα, Παρόλο που ήταν πολύ καλή η συνεργασία, φαντάζεστε ότι δεν συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία. Δεν τα καταφέραμε. Και θα κάνουμε και οι δύο προσωπικές τροπολογίες ως εισηγητές, αλλά αυτό δεν ε, αναιρεί καθόλου την κοινή προσπάθεια και την πρότασή μας. Α, γεια σου Κέι, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω ευχαριστίες της είπα την αποσία σου. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι μαζί σου. Τα βασικά στοιχεία λοιπόν ε, που συμμεριζόμαστε. Βασικό στόχο η προστασία, ενισχυμένη προστασία και αξιόπιστη προστασία των φορολογουμένων, όχι μόνο θεωρητική. Εξασφαλίζοντας και τη συστημική σταθερότητα ή επαναφέροντας τη σταθερότητα αυτή. Δεύτερος στόχος, να ενισχυθεί ταυτόχρονα και το θεσμικό πλαίσιο κατά την ανάκαμψη και εξηγένση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και εκ των προτέρων, αλλά και αυτή τη στιγμή ξεσπάσει η κρίση. Τι κάναμε λοιπόν, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ανάκαμψη, δηλαδή να δώσουμε καλύτερα κίνητρα το πρώτο και σημαντικότερο σημείο είναι ότι τα σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει να είναι πιο δεσμευτικά. Στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατά τα άλλα ήταν εξαιρετική βάση για την εργασία μας, αλλά προσπαθήσαμε να τη βελτιώσουμε κατά κάποιο τρόπο, ε, θεωρήσαμε ή αισθανθήκαμε ότι θα ήταν καλύτερο Σε περίπτωση που κάποιος κεντρικός αντισυμβαλόμενος ε, θέλει να αποστεί της αρχικής πρότασης ανάκαμψη, όχι απλώς να το κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή όπως ήδη ισχύει, αλλά να ε, ζητεί και την άδεια να αποκλίνει. Και είναι από εκεί και πέρα θέμα οργάνωσης να ε, χορηγείται γρήγορα η άδεια αυτή, να εγκρίνεται το αίτημά του ή να απορρίπτεται με ταχύς ρυθμούς πάντα από την αρμόδια αρχή. Άρα, να είναι πιο δεσμευτική αυτή η προσπάθεια, ήταν ο βασικός μας στόχος και δεύτερος. Είναι ε, να, ε, όταν έχεις μια ανάκαμψη ε, υπάρχει μια απώλεια απορρόφησης. Δηλαδή είναι ε, δύσκολη η επιλογή και η επιλογή των μέσων που θα χρησιμοποιήσεις για το στάδιο της ανάκαμψης. Στη συνέχεια είχαμε το ζήτημα ε, των αποζημιώσεων. Κατά το στάδιο της ανάκαμψης θα πρέπει να προβλέπετε αποζημίωση σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος ε, επιζήσει, επιβιώσει. Το θέμα δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά και αμοιβαίου συμφέροντος. Δηλαδή έχουμε ε, το κεντρικό αντισυμβαλόμενο, έχουμε τον εκαθαριστή και ε, τους πελάτες και οι τρεις έχουν όφελος και έχουν και συμφέρον να υπάρξει η ανάκαμψη. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι απεριόριστη αυτή η αποζημίωση. γιατί κάποια στιγμή θα καταντήσει αυτός ο οργανισμός να μην είναι σε ε, διάσωση, σε επιβίωση, ούτε σε ε, καθαρίστη να είναι ένα είδος ζόμπι και οι μέτοχοι να ε, αναζητούν το αν έχει λόγο ύπαρξης διάσωσης ή όχι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε στο κείμενο, το νομικό κείμενο, ότι κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης δεν θα μπορούν οι μέτοχοι να αφαιρέσουν την ε, δυνατότητα απορρόφησης ε, των απολειών, δηλαδή να ε, επιτρέπουν να καταβάλλονται μερίσματα και μπόνους. Δώσαμε δηλαδή ε, στην πρόταση πολύ μεγαλύτερη δομή και διάρθρωση για το σκέλος της ανάκαμψης. Ε, δεν θελήσαμε μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες να αριθμίσουμε τα πάντα, γιατί υπάρχουν διάφορα είδη κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Σκεφτήκαμε τα διάφορα ε, συστήματα και σχέδια ανάκαμψης. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού μοντέλου. Τώρα για την εξυγίανση ε, είναι τελείως, μάλλον κάπως διαφορετική η κατάσταση. Εκεί υπάρχει μία αρχή που εξηγεί ε, τον αντισυμβαλόμενο και ε, ασχολείται με δύο πράγματα. Πρώτον, τη συστημική σταθερότητα και το δεύτερο, την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Να υπάρχουν λοιπόν ασφαλιστικές δικλείδες και να είναι πολύ πιο δύσκολο οι ιδιώτες να αμφισβητούν, να προσβάλλουν αποφάσεις της δημόσιας αρχής. και κατά τη διάρκεια ε, αυτής ε, της εξηγίασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, διάφορες βασικές αρχές για την απορρόφηση των απολειών και για την συνέχεια. Ξέρω ότι μακρηγόρησα, αλλά έχουμε αρκετά γενναιόδορη κατανομή του χρόνου για την έκθεση αυτή. Θέλω να πω δύο λόγια για όλη αυτή την αρχιτεκτονική του ΕΜΙΡ και έχουμε και ε, την ε, αναθεώρηση που επίκειται. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα και με το ενδεχόμενο του Brexit έχουμε το εξής, η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα είναι στην ενιαία εποπτεία Γιατί σε περίοδους κρίσης κινδυνεύει να ε, μην μπορεί να λειτουργεί και ταυτόχρονα έχουμε την ίδια ε, προσέγγιση για τους μεγάλους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αρχή εποπτική και εξυγίανση σε ένα νέο πλαίσιο, γιατί τώρα είναι λίγο άδικο το σύστημα και όταν μπαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα και περιπλέκονται. Ξέρω γιατί ε, θέλει να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα λειτουργούσε αυτό το σύστημα σε περίοδους κρίσης, ούτε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να δράσει απέναντι σε τρίτες χώρες όπου θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη εποπτεία σε περίπτωση ετεροδικίας. Δηλαδή είναι ένα είδος χωριού ποτέμκιν που έχεις μόνο το σκηνικό και δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο την εποπτεία, αλλά και το θέμα της ε, ε, ανάκαμψης και της εξυγένσης και της ε, κεντρικής αρχής. Και όπως κάναμε και στην Τραπεζική Ένωση, τίθεται το ερώτημα τι δημοσιονομική ικανότητα, πόσα χρήματα θα έχουμε στη διάθεσή μας για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι δύσκολο να ε, καταλάβουμε ή να δεχτούν τα κράτη-μέλη να υπάρχει ένας ενιαίος κεντρικός ε, μηχανισμός ή μια αρχή να, ε, και ενώ στη συνέχεια να τους δουν να πληρώσουν εκείνα τα σπασμένα. Για τις τροπολογίες, μία από τις τροπολογίες μου θα είναι μια πρόταση να δημιουργηθεί, να συσταθεί ένα ταμείο ενιαίο ταμείο ε, εξυγίασης για τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους, γιατί είναι προϋπόθεση αυτό. Να προχωρήσουμε προς την ενιαία ε, εποπτεία και μια αρχιτεκτονική για την ανάκαμψη και την εξυγίαση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάκοπ. Και τώρα η δεύτερη συνεισηγήτρια, η Κέι Σουίμπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και Γιάκοπ που ανέλαβες εσύ. Έτρεχα από την άλλη άκρη του κτηρίου και σε ευχαριστώ και για την συνεργασία που είχαμε τους τελευταίους μήνες και δεν είχα ξαναεργαστεί ως συνεισηγητής και δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο περίμενα λόγω ακριβώς της δικής σου συνεργασίας και του ότι αναγνωρίσαμε το ποιες ήταν οι διαφορές και σε ευχαριστώ. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ξεκάθαρο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την ανάκαμψη και εξυγίανση συστημικά σημαντικών σημείων της υποδομής της αγοράς και να μπουν αυτά σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα είναι το τελευταίο πλαίσιο και τελικά η εκαθάριση θα είναι το τελευταίο κομμάτι που θα ξεκαθαρίσουν οι G20 στο Pittsburgh το 2019. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα που δεν πρέπει να καθυστερήσει και δεν θα πρέπει επίσης να συγχέεται με τους πιο πολιτικούς φακέλους που αφορούν ακριβώς τα θέματα εκαθάρισης το διεθνέ πλαίσιο κεντρικών αντισυμβαλωμένων και αμοιβαιοποίηση του κινδύνου σημαίνει πως ε, τα μέσα αυτά είναι πλέον παγκόσμια. Το σχέδιο αυτό έκθεσης ε, συμμορφώνεται με τις εργασίες της σχετικής επιτροπής. Και όσον αφορά την ανάκαμψη και την εξυγίανση, απαιτείται νομική βεβαιότητα και διαφάνεια. Το σχέδιο έκθεσης προσπαθεί να τα ενισχύσει αυτά έτσι ώστε όλοι οι δρόντες των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται ή τι μέγεθος έχουν, θα έχουν μια δίκαιη μεταχείριση σε όλες τις φάσεις. Και σημασία έχει βεβαίως η προστασία των επενδυτών. Και αυτό θα γίνει μέσω της ευθυγράμμισης των κινήτρων, έτσι ώστε όλοι να θέλουν να υπάρχει ανθεκτικότητα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, έτσι ώστε αν συμβεί ο Αρμαγεδόν να υπάρχει η βεβαιότητα αλλά και η απαραίτητη ευελιξία. Και εδώ πέρα στο σχέδιο έκθεσης υπάρχουν κάποιες δικλίδες ασφαλείας, ε, κυρίως όσον αφορά την χρήση των χρημάτων των πελατών. Παραδείγματο χάρη, η χρήση των οριακών κερδών επιτρέπεται μόνο αφού έχει κριθεί αποτελεσματικό και έχει εξαντληθεί κάθε άλλη εναλλακτική. Και βεβαίως ε, κοιτάμε να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο θα επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως η πολυπλοκότητα αυτών των υποδομών της αγοράς σημαίνει πως ε, το να βλέπουμε την ανάκαμψη και την εξυγένση ως ένα σύνεχες είναι το κάτι το χρήσιμο. Αλλά βεβαίως ε, βλέποντας ακριβώς αυτή την μετακίνηση από την ανάκαμψη στην εξυγίανση ως ένα συνεχές είναι κάτι το οποίο μπορεί να παραλυφθεί αν η σχετική αρχή κρίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό και θέλει να προχωρήσει σε εξυγίανση. Και εδώ πέρα βεβαίως αναμένω και τις τροπολογίες των συναδέλφων. Από την φύση τους οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι έχουν και συμβιβάζουν διάφορα συμφέροντα, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όμως, σε περιπτώσεις αναταραχής της αγοράς, προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια σαφής ιεραρχία για να λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις. Ε, θεωρήσαμε ότι είναι, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ κατάστασης χρεοκοπίας και μη. Και όπου θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται κάποια διάκριση είναι η αρχή του κανείς πιστωτής να μην βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα πρέπει να οριστεί σωστά για να μπορεί να σταθεί σε δικαστήριο. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει οι αρχές της εξυγένσης να μπορούν να δρουν, αλλά θα έχουν ακριβώς μια τέτοια ξεκάθαρη και αυστηρή αρχή για να μπορούν να δρουν χωρίς επιφυλάξεις, γνωρίζοντας ότι αργότερα θα μπορούν να υπερασπιστούν τα όσα έκαναν. Ακριβώς το να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ ανάκαμψης και εξυγίασης έχει μεγάλη σημασία. Έχουμε λοιπόν μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας, προβλέπουμε και επιπλέον κεφάλαιο από τους συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες στιγμές, ενημέρωση των πελατών όπως και την ανάγκη αποζημίωσης των συμμετεχόντων για να βοηθηθεί η ανάκαμψη ενός κεντρικού αντισυμβαλωμένου για να εφαρμοστεί αυτή η αρχή του ουδής επενδυτής δεν θα βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα. Πρόκειται λοιπόν για μια συνολική απάντηση σε μια καλή πρόταση της Κομισιόν και αναμένω τη συνεργασία με τους κοιοδησηγητές για να την βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ανέκαμψες πάρα πολύ καλά και αυτό είναι άμα έχει κανείς σχέδιο ανάκαμψης. Το σχέδιό μας τώρα είναι 5 λεπτά για κάθε σκιώδη και προειδοποιώ την Κομισιόν ότι και εσείς θα λάβετε τον λόγο αν το θέλετε. Η Ντανούτα Χούμπνερ πρώτη από το ΕΛΚ, την οποία αντικαθιστεί ο Μπραιν Χέις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, δεν είμαι η Ντανούτα Χούμπνερ όπως βλέπετε, όμως... άμεσα Ευχαριστώ. Όχι απλώς ε, λάθος κουμπί. Η Ντανούτα ζητά από τους δύο συνεισηγητές να, την να τη συγχωρούν, αλλά θα συνεχίσει τη συνεργασία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μαζί σας. Καλωσορίζει το σχέδιο της έκθεσης που φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στο κείμενο της Επιτροπής που ήταν μια σταθερή βάση, ένα καλό σημείο αφετηρίας. Αυτό που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι τα τέσσερα βασικά σημεία που ε, μπόρεσαν οι εισηγητές να χρησιμοποιήσουν ως απάντηση στα, στις του ΕΛΚ. Περισσότερη σαφήνεια για τα σχέδια ανάκαμψης, στην πρόταση της Επιτροπής δεν υπήρχαν αρκετές λεπτομέρειες, οπότε υπήρχε πολύ περιθώριο οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι να αποκλίνουν από τα σχέδια ανάκαμψης αυτής. Τώρα υπάρχει περαιτέρω ε, διαλεκτικότητα και το ζήτημα αυτό έχει επιληθεί. Μεγαλύτερη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα για τους πελάτες και τα μέλη, οι συνεισηγητές, την ε, ακολούθησαν αυτή την προσέγγιση από την αρχή και από τις συνομιλίες μας, τις συναντήσεις των σκιωδών, βλέπουμε ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να στηριχθεί από όλη τη διαγματευτική ομάδα. Δεύτερον, περαιτέρω διαφάνεια για τα σχέδια ανάκαμψη για τους πελάτε και τα μέλη. Εδώ βλέπουμε ένα σαφέ χάσμα σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Υπήρχε πολύ μεγάλο περιθώριο για το πώ θα δημιουργείται διαφάνεια προς τους πελάτες και τα μέλη για το ποιοι θα συμμετέχουν και θα σχεδιάζουν τα σχέδια ανάκαμψη. Τώρα ε, αναζητούμε επιπλέον τρόπους για να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια, ενώ η απόφαση της κατέρνηση που, αναλαμβάνεται, ε, που αναλήφθηκε εδώ είναι πρόσδεκτη. Επίση, το να ε, προστατεύονται τα χρήματα των φορολογουμένων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι συνεισηγητέ ήταν πολύ σαφεί για το θέμα αυτό ευθύ εξ αρχή. Του υποστηρίζουμε και σε αυτό το σημείο επίση, και βάσει των συζητήσεων που κάναμε ω τώρα, ελπίζουμε ότι η Δημοκρατική Ομάδα θα παραμείνει ενωμένη. Επίση, είμαστε ικανοποιημένοι που οι συνεισηγητέ ακολουθούν την κατεύθυνση τη καλύτερη ε, αποσαφήνιση των σεναρίων πτώχευση και μη πτώχευση. Χρειάζεται αυτή η διευκρίνηση για, την, ε, για τον καθορισμό τη οικονομική συμμετοχή του κεντρικού αντασυμβελωμένου ανάλογα με το κάθε σενάριο που θα ισχύει. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση και είμαστε της άποψης ότι αυτή η διαφορά που έχει οριστεί πρέπει να ξεκαθαριστεί με μεγάλη σαφήνεια και στις δύο περιπτώσεις. Πτώχευση και πτώχευση. Κατά τα άλλα έχουμε κάποιε αμφιβολίε για την προσέγγιση της έκθεση σε τρει τομεί. Πρώτον, το θέμα του νέου άρθρου 20α που έχει να κάνει με τις αποζημιώσει για την ανακαμψή και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι πελάτε ή οι μέλη και ενώ συμμεριζόμαστε το στόχο των συνεισηγητών και εγκρίνουμε τη Γενική Αρχή έχουμε ακόμη αμφιβολίε για τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα θα λειτουργεί ε, με τον τρόπο που περιγράφεται στην έκθεση τώρα. Συγκεκριμένα ο αριθμός που προτείνεται ε, είναι περί τη λεπτομέρεια και θα έπρεπε απλώς να ακολουθήσουμε τη γενική αρχή. Επίσης, ε, το θέμα του No Creditor of ε, και η σχετική αρχή στην τωρινή της διατύπωση. Πρέπει να κοιτάξουμε να υπάρχει προσέγγιση με την αρχή του FSB για μια καλύτερα συντονισμένη προσέγγιση γενικώ, αλλά και σε σχέση με το κόστος που έχει εντοπιστεί ως προβληματικό, είναι κατανοητό ότι από θεωρητική τουλάχιστον άποψη θα προκύψουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Και έπειτα έχουμε ανησυχίες σε σχέση με το Ταμείο εξυγίανση, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι βλέπουν με συμπάθεια οι συνεισηγητέ. αλλά φαίνεται ότι δεν θα είναι απλό, δεν θα είναι να έχουμε ένα τόσο, τόσο γρήγορα ένα ταμείο στο και μικρό. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε πολύ ρευστότητα και το κόστος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο καθώ είναι χρήμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλου σκοπού. Τέλο, για τα θεσμικά ζητήματα, για τα οποία καταλαβαίνω ότι προς το δεν υπάρχει συμφωνία στην έκθεση. Είμαστε υπέρ μιας ευρωπαϊκότερης προσέγγισης στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Και αυτό θα μπορούσε περαιτέρω να διευκριστεί στην έκθεση ΕΜΕΡΔΙΟ. Το σύστημα εποπτείας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση συνολικής ανακαίνησης. Οπότε, ε, καθώς δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αυτό που θέλουμε να βεβαιωθούμε είναι ότι η προσέγγιση της εποπτείας θα προβλεφθεί στο τελικό οικοδόμημα. Άρα, κατά την άποψή μας, είναι πρόημο να οριστεί στο κείμενο μια νέα αρχή εξηγήσεως πρέπει να συμβαδίσει αυτό το σχέδιο με τα υπόλοιπα όσα εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Και κάποια θεσμικά ζητήματα μπορούν να επιληθούν, αλλά δεν είναι ανάγκη να μείνουν και τελείως ασχεδίαστα λόγω ενός από αυτά. Α αφήσουμε λοιπόν μια ρήτρα με ένα επαρκέ χρονικό διάστημα, ώστε να επιληθούν και οι υπόλοιπε θεσμικέ διευθυντήσει για το θέμα τη εξυγίανση και έτσι να μπορέσει να προσαρμοστεί και αυτό που τώρα βλέπουμε. Δηλαδή να φροντίσουμε να υπάρξει συνοχή ε, μέσα στο διάστημα εντό του οποίου θα εγκαθιδρυθεί αυτή η ενιαία αρχή εξυγίανση. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να εργαστούμε καλύτερα όταν θα έρθει αυτή η στιγμή. Σε ευχαριστούμε, Μπράιαν. Για την άλλη, κυρία Φανούβεν Χόζεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω με ευχαριστίες προς τους δύο συνεισηγητάς. Όπως είπε και ο Γιάκοπ Φον Βάιτσέκερ, ε, είναι ένα παράξενο ζευγάρι αυτό, δύο εισηγητές, ο ένας από το, η μία από το ΙΣΙΑΡ και ο άλλος σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ξέρουμε ότι δεν είναι γάμος από έρωτα, αλλά τα προξενιά καμιά φορά διαρκούν περισσότερο γιατί δεν βασίζονται τόσο στο συνέστημα όσο στη λογική και για μια νομοθετική έκθεση αυτό δεν είναι και τόσο κακό θα έλεγα. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι ότι ε, είναι λογικά όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους και μας ενώνουν και όπως είπε και η ΚΕΙ ε, υπήρξε μια καλή βάση πρώτα Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και οι δυο σας κάνατε Πολύ καλή δουλειά, το βελτιώσατε πάρα πολύ το αρχικό κείμενο. Είναι σημαντικό το, τμήμα αυτό. Ε, λείπει από το, την νομοθεσία για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Και για μας είναι σημαντικό να προσαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με τη, διεθνώς ισχύοντα. Ε, γιατί ξέρουμε ότι το clearing είναι καταξοχήν διασυνοριακή ε, ε, δραστηριότητα. Λοιπόν, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά συμφωνώ και με τα όσα είπε ο συνάδελφος Μπράιν Χέις, εξ ονόματος της Δανούτα Χιούμπνερ. Υπάρχουν μερικά σημεία που χρειάζονται κάποιο χτένισμα. Ε, θα αναφερθώ σε αυτά τα τρία. Μια που άρχισε τη συζήτηση ο Γιάκοβ ε, για το ενιαίο μηχανισμό ή το ενιαίο ταμείο εξηγένσης. εμείς δεν θα θέλαμε να το ανακατέψουμε τώρα σε αυτό το ζήτημα, σε αυτό το θέμα. Το θέμα που μας απασχολεί είναι πολύ τεχνικό, ας το κρατήσουμε έτσι λιτό και περιορισμένο και σε λογικά πλαίσια, γιατί αν μπούμε τώρα στις πολιτικές συζητήσεις που κρύβονται από πίσω, καήκαμε. Αυτό καλύτερα δηλαδή να το κάνουμε στην αναθεώρηση ε, και Mir, γιατί υπάρχει κίνδυνος στο συγκεκριμένο θέμα να το καθυστερήσουμε αν μπούμε σε τέτοια ε, ζητήματα και θα ήταν κρίμα. Για τα θέματα της απώλειας ε, στην ανάκαμψη σε περίπτωση μη πτώχευσης ε, προτείνουν οι συντονιστές να μην το θίξουμε αυτό και να μεταφερθεί στους αντισαβαλωμένους και στους μετόχους. Βεβαίως, για να περιορίσουμε ε, τους κινδύνους και να εξασφαλίσουμε την ε, σταθερότητα ε, και την ποικιλομορφία στους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους. Εδώ είναι μια λεπτή ισορροπία όπου πρέπει να βρεθεί ανάμεσα στα δύο. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα τι ακριβώς θέλουμε με χαρά να το συζητήσουμε στη συνεδρία των σχεδόν ε, εισηγητών πρώτη είναι αύριο. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά ε, τη, τους ορισμούς στα θέματα του. Κανένας πιστωτής να μην είναι σε χειρότερη μοίρα. Ε, ξέρουμε ότι ο διάβολος λέμε, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ένας ε, πολύ περιοριστικός ορισμός, πολύ στενός ε, θα μπορούσε να περιορίσει πολύ την ε, δραστηριότητα μιας αρχής, αλλά ήταν πάρα πολύ ευρύ ο κανονισμός, μάλλον ο ορισμός, ε, τότε θα υπάρχει δυσκολία συγκεκριμένων υπολογισμών ε, σε περιπτώσεις κρίσης και θερμό. Αυτά θα δούμε τις ερχόμενες εβδομάδες. Και τρίτον, ένας βασικός στόχος του νομοθετήματος αυτού είναι η προστασία των δημοσίων χρημάτων. Αλλά μην δώσουμε λάθος μηνύματα για να μην αυξήσουμε τον ηθικό κίνδυνο. Να μην λοιπόν ε, κάνουμε προτάσεις που μπορεί να δίνουν κίνητρα για ένα bail-in για τη διάσωση ε, των αντισυμβαλωμένων. Ε, Με χαρά να συνεργαστώ μαζί στις επόμενες εβδομάδες και προσβλέπω στη συνεργασία αυτή για περαιτέρω βελτίωση του φακέλου. Ευχαριστώ κόρα και και το χρόνο σου απολύτως. Από την ΚΟΟ, ο κύριος Βιέγας, για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ο κανονισμός αυτός παραδοσιακά είναι και σε αυτούς που μας δυσκολεύουν να σχολιάσουμε. Μιλάμε για ίδρυση θεσμών που κατευθύνουν την οικονομία σε αντιδιαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που εμείς ε, ευαγγελιζόμαστε με το δικό μας οικονομικό μοντέλο. Ουσιαστικά γίνεται το παν η χρηματοπιστωτική διάσταση της οικονομίας και αυτό επιβαρύνει τα ίδια τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν στον τομέα αυτό. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που λέει ότι θέλει να επιφέρει σταθερότητα για τους διάφορους παράγοντες της οικονομίας. Καταλήγουμε να δημιουργούμε πηγές ε, διακυμάνσεων, αναταράξεων και αστάθειας. Αυτές οι κεντρικές αρχές, οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι, οι οποίοι αρχικά δημιουργήθηκαν για σκοπούς αποτελεσματικότητας και το καθεξής, τελικά γίνονται ένας επιπλέον παράγοντας συστημικού κινδύνου δημιουργούν επιπλέον αρχές, φορείς ε, μεγάλων διαστάσεων ε, προκειμένου να πτωχεύσουν. Και έχουμε πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τραγωνισμού του κύκλου. Θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο. Μόνος τρόπος να μειώσουμε τον κίνδυνο είναι να υπάρξει μεγαλύτερη κλίμακα και τελικά αυτό προκαλεί κινδύνους συστημικούς με θεσμούς που είναι too big to fail. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σε μια, μπροστά σε μια κατάσταση όπου εμείς δεν αναγνωρίζουμε τους δικούς μας στόχους και τις δικές μας ιδεολογικές αρχές. Καταλαβαίνουμε το θέμα, καταλαβαίνουμε την ανάγκη να ρυθμιστούν οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι και υπ' αυτήν την έννοια Δεχόμαστε το μεγαλύτερο μέρο της έκθεσης. Βέβαια, σε περίπτωση πτώχευση ε, μιας τέτοια, ε, η περίπτωση πτώχευσης μιας τέτοιας αρχής, του κεντρικού αντισυμβαλόμενου είναι μικρή. Αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει πρόβλεψη και για να ελαχιστοποιηθεί αυτό ο κίνδυνο όσο και αν είναι ήδη μικρό. Γι' αυτό λοιπόν και με όλε τι κρίσιμε ε, τυχαίε και παρατηρήσει που καλύπτει η έκθεση, εκεί τα λαμβάνουμε υπόψη. Πρέπει να μειωθεί η περιπλοκότητα. Το θέμα της ιδιοκτησίας των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, το μοντέλο διαχείρισής τους, όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα δούμε και ακόμη πιο ε, αυστηρά. Ε, δηλαδή, το μοντέλο διακυβέρνησης να περιοριστεί μόνο σε μερικά χρηματοπιστωτικά ενεργητικά που τα διαχειρίζονται αυτοί οι αντισυμβαλόμενοι σε πολύ συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, αυτά που είναι τα πιο επικίνδυνα, ίσως ήταν τα μόνα που θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης για να μειωθεί η δυνατότητα η περίπτωση διακυμάνσεων και κινδύνων. Και εδώ πρέπει να βρει το κατάλληλο σημείο ισορροπία μεταξύ των αυστηρών άκαμπτων κανόνων και τη ελαστικότητα, τη διαλλακτικότητα που χρειάζεται για να μπορέσουν αυτοί οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι να διαχειριστούν τι υποθέσει τους και αν χρειαστεί να παρέμβει ο επόπτης, ο βλέπουν. Πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Και επί της ουσίας, αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο σήμερα και πρέπει να υπογραμμιστεί, το δεχόμαστε. Δηλαδή πρέπει οι ευθύνε των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και όσοι ενεργοποιούνται στην αγορά πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να προστατευθούν, να ε, γλιτώσουν οι φορολογούμενοι. Επίσης για τα ταμεία αντασφάλισης, αλληλασφάλισης μάλλον, και κυρίως ό,τι αφορά την επιστημιστική ασφάλεια, θεωρούμε ότι και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με την φυσική αυτή παρατήρηση ότι είμαστε σκεπτικιστές από την άποψή μας και από τη δική μας σκοπιά καμία προσπάθεια διακανονισμού και ε, διευθέτησης δεν μπορεί να απλοποιήσει το ρόλο αυτών των κεντρικών αντισυμβολωμένων. Θα συμβεί το ίδιο που συνέβη και με το ενίο Ταμείο Εξυγένσης, με την Τραπεζική Ένωση. Σήμερα βλέπουμε ότι είναι ανεπαρκές και ότι υπάρχει επιτάπητο η ανάγκη να δημιουργηθεί μηχανισμός ο οποίος θα αναθεωρήσει όλο αυτό το οικοδόμημα. Κάτι ανάλογο θα γίνει και εδώ. Όλες αυτές οι λύσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες, αλλά θα κλείσω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Τα προβλήματα υπάρχουν, εδώ καλούμαστε να τα λύσουμε στην πράξη. Γι' αυτό λόγω της φύσης της έκθεσης καταλαβαίνουμε και την ανάγκη να ρυθμιστούν αυτά τα θεσμικά όργανα, αυτές οι, μάλλον οι αρχές, οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι, οι οποίοι αφού δημιουργήθηκαν κινδυνεύουν να γίνουν παράγοντες αστυνομικού κινδύνου και αυτό θέλουμε και να προλάβουμε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε τελευταίος, τελευταία μάλλον από τους Πρασίνους η κυρία Μόλι Σκοτ Κάτω. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα σχολάσω την σχέση μεταξύ των συνσηγητών. Θα προκύψει αυτό στις συζητήσεις. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως θεωρούμε εμείς ότι εμείς οι πράσινοι ότι βελτιώνουν το κείμενο της Κομισιόν και θα διευκολύνουν έτσι τη δουλειά μας ημών των σχεδόν συγκητών. Επίσης, βεβαίως, συμφωνούμε με την έμφαση του ότι θα πρέπει να, να διανέμονται οι ζημίε ανάλογα με το πώ ο καθένα μπορεί να αξιολογήσει του κινδύνου να κεντρικών αντισυμβαλωμένων και να αναλάβει τα κατάλληλα βήματα και βεβαίω να υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ χρεοκοπία και μη. Μα αρέσει το ότι οι εισηγητέ σκοπεύουν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια στην ιεραρχία των ε, ζημιών. Επίσης θεωρούμε ότι το βάρος ε, της ε, αποδείξεως να πέφτει σε όσους θέλουν να εμποδίσουν την εξυγένση είναι σωστό και βεβαίως η σοφία εκ των υστέρων δεν μετράει πάρα πολύ και τέλος είναι θετικό το ότι ξεκαθαρίζει ότι η εξυγίανση βεβαίω είναι μια ανησυχία η οποία δεν υφίσταται όταν έχει ήδη κλείσει ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος. Κάτι το οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε με τους σκιώδει είναι το εξή. Πρώτα απ' όλα σύμφωνα με την τροπολογία 86, σε περιπτώσει μη χρεοκοπία, ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος έχει τρεις φορές περισσότερο ίδιο συμφέρον σε σχέση με την χρεοκοπία αμφισβητούμε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεδομένου του ότι τα μέλη του μηχανισμού εκαθάρισης είναι επίσης μέλη της Σχετικής Επιτροπής. Επίσης, ε, τα ανοίγματα σε μετρητά που αναφέρονται στο Πολυγείο 87 ε, αφορούν ή όχι το κεφάλαιο του κεντρικού αντισυμβαλωμένου. Και τέλος θα πρέπει ο ορισμός χαροκοπίας και μήνα ευθυγραμμιστεί με τροπολογία 83. Στην τροπολογία 51 θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία της εξυγένσης από τις άλλες ε, λειτουργίες ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει γενικώ μεγαλύτερη ανεξαρτησία από ό,τι προτείνεται το σχέδιο έκθεση. Οπότε οι τροπολογίε μα θα εστιάσουν σε λίγα από τα ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν την πρόταση. Πρώτα απ' όλα, οι στοχευμένε εξαιρέσει για τι κεντρικέ ε, τράπεζε ε, και τι ε, κρατικές υπηρεσίες χρέους για οποιοδήποτε μπέιλιν. θέλω να τονίσουμε τον ρόλο της ΕΣΜΑ. Μια πιθανή αντικατάσταση του κειμένου του επίπεδου 1 με κάποιες τεχνικές προδιαγραφές για να υπάρξει η δυνατότητα ρυθμίσεων υπό το φως της εμπειρίας, μία απέτηση για το εάν τα μέσα κρατικής χρηματοδότησης ως última ratio σημαίνουν ότι χρειάζονται κρατικά λεφτά και τέλος θα θέλαμε να εισαχθεί μια απέτηση η κεντρική αντισυμβαλόμενοι να χρησιμοποιούν τεχνολογία σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ε, με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει στα stress test αυτά και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Σύντομο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στο ΚΕΤΣΙΑ, να ρωτήσω την Κομισιόν, τον κύριο Πίρσον, να μας πει δύο λόγια. Να σας πω τρία, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που Εκτιμάται ε, ότι είναι καλή βάση νομοθετική μας πρόταση. Ε, δεύτερο σχόλιο. Καμία από τις τροπολογίες που προτείνονται δεν ε, είναι προβληματικές και θα συστήσουμε στο Συμβούλιο με χαρά να προχωρήσει στη συζήτηση αυτών των προτάσεων. Θεωρούμε όλες τις προτάσεις σας συνιστούν βελτίωση στην αρχική δική μας και ε, καλωσορίζουμε και τις τροπολογίες των εισηγητών που ζητούν πιο δεσμευτικές ε, ρυθμίσεις. Το θέμα είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί σε περίπτωση κρίσης ε, όλο αυτό το σύστημα ανάλογα με το τι ισχύει σε περιπτώσεις πτώχευση μη, ε, ανάκαμψη και εξυγίαση, Όλες αυτές οι προτάσεις είναι πάρα πολύ ε, λογικές και σύμφωνα με τις ε, διεθνώς ισχύους διατάξεις, ε, όχι σε μερίσματα, όχι σε βόνους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικά και για την προστασία των φορολογουμένων και για την προστασία των πιστωτών και των επενδυτών. Γενικά είναι εξαιρετικά καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση. Ένα τελευταίο σε σχέση με τα όσα είπε ο συνεισηγητής κύριος Φων Βάιτσέκερ. Ενδιαφέρον αυτό που πρότεινε. Στη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το εξετάσαμε αυτό το θέμα του Ταμείου για την Εξυγένση για πέρσι το Νοέμβριο, αλλά δεν επιλέξαμε αυτή τη λύση. Υπήρχε για, για τις τράπεζες αυτό το σύστημα 44,3 δισεκατομμύρια δίνουν τα κράτη-μέλη και επίσης για τους αντισυμβαλωμένους. Αν καταλαβαίνω καλά αυτό που προτείνει ο συνεισηγητής είναι να σκεφτούμε να υπάρξει ένα τρίτο ταμείο ε, για την εκαθάριση. Αναφέρουμε στην αξιολόγηση μας και τη μελέτη αντικτύπου. Κατανοώ τα όσα λέει ο, ο εισηγητής και από τις ε, αντιδράσεις ότι δεν είναι μια μεμονωμένη ιδέα ε, να το συζητήσουμε, είπε στο Κοινοβούλιο, το θέμα της ίδρυσης ενός ταμείου. Αλλά εδώ πρόκειται για θέματα δημοσιονομικής ευθύνης. Ε, καλωσορίζουμε την ανάγκη συζήτησης που ε, έθεσε ο εισηγητής, αλλά εδώ έχει σημασία και η χρονική ακολουθία. Το ταμείο είναι η απόρρεια μιας αρχής ε, εξυγίανσης ενιαίας και αυτό απορρέει από την ενιαία αρχή ε, εποπτείας. Άρα πρώτα θα δούμε την κοινή εποπτεία, μετά θα δούμε την κοινή εξυγίανση και στο τέλος την κοινή ενιαία ε, χρηματοδότηση όλων αυτών. Πάντως ε, είναι καλό που έθεσε αυτό το θέμα τουλάχιστον εισηγητής προς συζήτηση για το Ταμείο Εξηγένσης. Θα δούμε όμως ποιο πρέπει να γίνει πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Αυτά Πρόεδρε και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε τη Η κυρία Μπερές πρώτη. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω Εάν ο γάμος αυτό βασίζεται στον ορθολογισμό, τόσο το καλύτερο αν έτσι είναι. Αλλά για την πρόταση των εισηγητών, ήθελα να αναφέρω και εγώ δύο-τρία από τα θέματα που μα ανησυχούν. Πρώτα απ' όλα, είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση και καλώ ήρθε στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί ο τρόπο που Ξηγαίνουμε τα της οικονομικής κρίσης από 2008 έχει δημιουργήσει νέους κινδύνους για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι ε, έχουν γίνει και το παραδέχεται και η διεθνής κοινότητα πιο συστημική από ήταν πριν. Ή τέλο πάντων συστημική με διαστάσεις σημαντικότερες από ό,τι στο παρελθόν. Είμαστε σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στις χρηματαγορές και είναι η καταλληλότερη στιγμή για να δούμε και κατεπηγόντως μάλιστα τον συστημικό κίνδυνο που αυτή τη στιγμή ενέχουν οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει στην εξέταση αυτής της έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι τα πάντα μπορεί να βρίσκονται σε κάθε σημείο του συστήματος, αλλά εμείς πρέπει να πάρουμε το σωστό σημείο του παρατηρητή, ε, το σωστή τοποθέτηση και να εντοπίσουμε αυτό το κουβάρι από πού θα το ξεμπλέξουμε. Γιατί δεν γίνεται όλα να είναι αλληλεξαρτώμενα μεταξύ τους μέχρι τέλους, διότι με την κατανομή του κινδύνου και την ανάληψη ευθύνης μπλοκάρουμε τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν συγκεκριμένε προτάσει. Τι θα κάνουμε, πώ θα βελτιώσουμε τα πράγματα δεδομένου του κινδύνου ε, και του κεντρικού αντισυμβαλωμένου, ποια θα είναι τα προγράμματα για την ανάκαμψη και για την εξυγίανση με πολύ συγκεκριμένου όρου, του οποίου πρέπει να του εξετάσουμε στο σημερινό πλαίσιο. Τώρα, αν ναι, εντωμεταξύ στο, στο μέλλον τα πράγματα αλλάξουν και χρειαστεί θεώρηση, θα το κάνουμε. Εάν, εάν περιμένουμε να ε, τελειοποιηθεί όλο το οικοδομικό, όλο το αρχιτεκτόνημα, το οικοδόμημα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Και μετά να τα προβλέψουμε όλα για να σκεφτούμε πώς θα διασώσουμε, πώς θα ανακάμψει και θα εξηγιανθεί ένα κεντρικό αντισυμβαλόμενο σήμερα, δεν θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Είναι ένας κίνδυνος που δεν χρειαζόμαστε. Δεύτερο στοιχείο για την εξισορρόπηση της ανάκαμψης και με την εξυγίανση. Καταλαβαίνω το στόχο των εισηγητών είναι να δώσουν περισσότερη έμφαση στη φάση της εξυγίανση. Διότι, μάλλον της ανάκαμψης, διότι ό,τι γίνει υπέρ τη ανάκαμψη και μας επιτρέψει να αποφύγουμε τα τη εξυγίανση είναι το, το καλύτερο. Η πρόταση αυτή δηλαδή δίνει κίνητρο στους εμπλεκομένους, τους φορείς, να πάνε και στην εξυγίανση αν χρειαστεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ε, διευκρινιστεί ή αν παραμένουν αποκλεισμένοι μόνο στο επίπεδο της ανάκαμψης. Και σε ό,τι αφορά το Ταμείο της Εξυγίανσης, το συζήτησα με τον συνάδελφο Βάιτσεκερ, ε, ξεκίνησε όλη η συζήτηση γιατί κάποιες τροπολογίες θα προκύψουν. Αλλά πρέπει να πω ευθύ εξ αρχή ότι για μένα το θέμα τη αναλογικότητα ενό τέτοιου ταμείου και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα είχε πει περισσότερε λεπτομέρειε αριθμητικέ. Τέλο πάντων, αυτό που του είπα είναι ότι αν θέλουμε ένα αξιόπιστο ταμείο εξηγιασίε θα πρέπει να φτάνει τα 500 δι ευρώ. Να ξέρουμε δηλαδή τι λέμε και να προσπαθήσουμε να είμαστε ακριβείς και αποτελεσματικοί για τα υποθετικά σενάρια του μέλλοντος. Εφόσον ε, κάτι γίνει και υπάρξει πτώχευση για το Ταμείο Ξηγένση, Τώρα για όλους τους ε, φορείς που συμμετέχουν εδώ. Γίνεται πολλής λόγος για τράπεζες, αλλά αν μιλάμε για μία δραστηριότητα αποζημίωσης, δεν είναι μόνο οι τράπεζες που εμπλέκονται. Ε, η πραγματικότητα των συναλλαγών μα φέρνει και άλλε αρχέ και παράγοντε υπόψη. Για να μην ξεχνάμε τη φύση και τον χαρακτήρα των κινδύνων που στοχεύουμε. Και να θυμίσω ότι κατά την επίσκεψη τη περασμένη εβδομάδα στην Washington με όσου ε, συζητήσαμε από την Αμερικα... συναντήσαμε από την Αμερικανική πλευρά ήταν όλοι σύμφωνοι λέγοντας ότι οι asset manager δεν αμφιβάλλουν για τη σημασία του θέματο, αλλά δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να είναι αυτοί υπεύθυνοι για την ε, ανάκαμψη των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Ευχαριστώ, δεν έχω δει κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Έτσι είναι. Εάν ναι, τότε θα ήθελα να στραφώ στους συνεισηγητές μας ε, με ναι, την αντίστροφη σειρά να ακούσουμε πρώτα την άποψη της Κέιτ και μετά τον κύριο Φων Βάστισεκερ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Δεδομένου του ότι έχουμε... είμαστε σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικοί, έχουμε ξεκινήσει από τις αντίθετες ε, πλευρές του φάσματος και κάπου στη μέση έπρεπε να συναντηθούμε. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε από αυτό και να παραμείνει ως τεχνικό θέμα θα πω το εξή. Προφανώς ε, έχουμε περάσει σε ζητήματα ενιαίας εποπτικής αρχής ε, και ταμείου εξυγένσης. Δεν υπάρχει στο κείμενο, θα φανούν αυτά στις ε, τροπολογίες, επειδή δεν συμφωνούμε ακριβώς από Νομίζω τα σχόλια του Γιάκομπο ότι Ε, περιλαμβάνεται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Μάλτας στον νέο υποπτικό μηχανισμό, ενώ όχι η κεντρική αντισυμβαλόμενη που είναι παγκόσμιες εταιρείε. Ε, να σας πω, ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό ήταν για να σπάσει ο δεσμός μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και η επιρροή που είχαν στο τραπεζικό σύστημα. Δεν έχει σχέση με το μέγεθος της εν λόγω τράπεζας. Οπότε, πρέπει να το πω αυτό, δεν φορά την ικανότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να εργαστεί και το Εποπτικό Συμβούλιο για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους από την εισαγωγή του ΕΜΗΡΙ το 2013 εργάζεται πάρα πολύ ικανοποιητικά και όλη η δουλειά η οποία γίνεται παγκοσμίω τώρα στο εποπτικό αυτό συμβούλιο ε, είναι αρκετά ικανοποιητική. Όταν μιλάμε για κεντρικού αντισυμβαλόμενους πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο ΕΜΗΡ ήταν πραγματικά το μέτρο σύγκρισης ε, για το πόσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και πλέον το μοντέλο ε, δουλεύει με τρόπο που δεν είχε ποτέ σχεδιαστεί προκρίσεις. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και θεωρώ ότι αν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό το θέμα από τα πιο πολιτικά ζητήματα που έχουν προτείνει πολλοί, τότε θα κάνουμε μια χάρη σε όλους. Γιατί όσο το συντομότερο έχουμε αυτά τα ζητήματα περί ανάκαμψης και εξηγένσης σε νομοθεσία θα είναι καλύτερο γιατί έτσι θα, θα συμπεριφέρονται όλοι όπως θα πρέπει σύμφωνα με την ιεραρχία της χρεοκοπίας. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε μια νομοθεσία εδώ πέρα που δεν θέλω να χρησιμοποιηθεί και αν την συντάξουμε σωστά δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φανβάιστσεκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Θα ξεκινήσω με εσάς κύριε Μπρέν. Ε, συμφωνώ με αρκετά από αυτά τα οποία είπατε. Υπάρχει μια πτυχή όπου θεωρώ ότι υποτιμούμε την σημασία αυτού του ζητήματος ε, του τι δηλαδή σημαίνει ικανότητα προφήσης ζημιών και εξυγίανση αυτή τη στιγμή. Γιατί βεβαίως ε, το θέμα είναι του πώς η κεντρική το πώς λειτουργεί η κεντρική τράπεζα. Γιατί εδώ πέρα βερβάνς κανείς δεν λέει ότι τα 500 δισεκατομμύρια ρευστότητα θα πρέπει να τα δώσει κανένα ταμείο, ούτε το λέει κανείς για το τραπεζικό σύστημα. Γνωρίζουμε πως ε, ένα ταμείο εξυγίανσης ε, τραπεζών θα είναι ανεπαρκές ε, και τα έχουμε πει πολλές φορές. Γι' αυτό χαίρομαι που το συζητάμε σε αυτήν την συγκυρία, την εμπλοκή δηλαδή των κεντρικών τραπεζών. Αλλά τότε έτσι ε, συζητάμε μέσως και την εμπλοκή των φορολογουμένων. Γιατί αυτοί σχετίζονται και συνδέονται με τις κεντρικές τράπεζες μέσω της εκταμίευσης ή των κερδών των κεντρικών τραπεζών. Οπότε ακόμα και σε μια κατάσταση εποπτική εποπτικής αρχής, η δυνατότητα απορρόφησης ζημιών σε περίπτωση εξυγένσης νομίζω πως είναι απολύτως σωστή. Γι' αυτό και πάλι, κόρα, συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία είπατε, αλλά υπάρχει ένας τομέα ε, τομέας όπου θα πρέπει να κάνουμε την διάκριση που κάνατε μεταξύ του πολιτικού και του λογικού. Πρώτα απ' όλα, ε, δεν είμαι σωστή. Δεν είμαι σίγουρο εάν τιμούμε την λογική όλων εδώ μέσα. Και δεύτερον, πρόκειται για μια λανθασμένη υπόθεση. Υπάρχει ένα πολύ υπαρκτό ερώτημα. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα ρωτήσουν τα κράτη-μέλη το τι σημαίνει και τα ποσά βεβαίω τα οποία εμπλέκονται. Σημαίνουν ότι η ε, πιθανότητα αυτή θα είναι μικρή. Αλλά αν δεν είχαμε εφεύρει την φράση πολύ μεγάλε για να χαρακοπήσουν, θα έπρεπε να έχουν εφευρεθεί για του κεντρικού αντισυμβαλόμενου πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε τράπεζα. Οπότε το θέμα του να μιλάμε για την δυνατότητα απορρόφηση ζημιών στην εξυγίανση είναι κάτι το ρεαλιστικό, γιατί βεβαίω πάντα μπορούμε να ε, ισοσκελίσουμε τον ισολογισμό εάν παραβιάζουμε τα συμβόλαια. Αλλά βεβαίω τότε επικρατεί μεγάλη αναταραχή και η πραγματική έννοια της, της έννοιας ε, απορρόφησης ε, ζημιών και εξυγίανσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Πολύ σοβαρά. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα της ε, μόλις για stress test των κεντρικών αντισυμβαλωμένων έφυγε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τις τα μεταφέρετε για να έχουμε έναν πιο επίσημο τέτοιο μηχανισμό. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, ε, μια πολύ θετική πρόταση. Και για αυτό το οποίο είπε ο Παρατεκπίρσεν, ναι, πράγματι, η σειρά προτεραιότητας έχει μεγάλη σημασία. Και συμφωνώ και βέβαια η πολιτική πτυχή θα ήταν διαφορετική. Και αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ίσως η Κομισιόν είχε προτείνει μια ακολουθία διαφορετική. Θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει με την μεταρρύθμιση της ε, ΕΖΑ κτλ. Αλλά αντιλαμβάνομαι πλήρω ε, αυτό το οποίο σημαίνει. Δεν παραπονιέμαι ότι έτσι έρχονται τα θέματα και έτσι τα προχωράτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λογικά πρέπει να ακολουθήσουμε την ακολουθία αυτή που πρότεινε η Κομισιόν. Είναι νομίζω απολύτως θέμητο διανοητικά να συνδέσουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα σήμερα, ότι πρέπει να καθυστερήσουμε κάποια πράγματα μέχρι να λυθούν όλα τα άλλα. Σαφώ δεν είναι αυτή η στρατηγική μα Ε, μου και ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιακόμπ. Ευχαριστώ την Επιτροπή, τα μέλη, ε, ε, τους Κιώδης, όλους τους εισηγητές. Πληροφορίες τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Προθέσουμε για την υποβολή των υπολογιών 25 Οκτωβρίου εκτός να φτάσει έτοιμα για παράταση. 20 Νοεμβρίου ε, θα είναι μέγιστη δυνατή παράταση. 7 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ και τον Ιανουάριο στην Ολομέλεια. Ε, κατά τα άλλα, ε, δεν θα κάνουμε διακοπή, περνάμε απευθεία στο σημείο 7 γιατί έχουν ενημερωθεί εγκαίρω οι σκιώδε και θα έρθουν. Πλαίσια προελοπτική αναδιάρθρωση, δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την ενίσχυση τη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αναδιάρθρωση, αφαιρεγκαιότητα και απαλλαγή. Εδώ ο συντάκτη τη νομοδότηση είναι ο κύριο Τσαμπόν από την Άλμπε. Λίγα λόγια πρώτα. Πρώτα απ' όλα ε, θελήσαμε να είμαστε συναρμόδια επιτροπή, δεν τα καταφέραμε. Η πρόταση προτάθηκε ως μέρος της δέσμης μέτρων για τις τράπεζες. Και αυτό το σύστημα της προληπτικής αναδιάρθρωσης είναι σημαντικό για τις τράπεζες που έχουν ε, προβλήματα στα ισοζύγια τους και κόκκινα δάνεια. Έχουμε 278 τροπολογίες και ετοιμάζονται συμβαστικές τροπολογίες σε πολλούς τομείς. Να περάσουμε απευθείας λοιπόν στη συζήτηση και ο κύριος Τσαμπόν έχει πέντε λεπτά για την εισήγησή του, μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπους εισηγητές, ΚΑΤΔΙΑ, η Επιτροπή κτλ. Κύριε Τσαμπόν, αν είστε έτοιμος. Πανέτοιμος, ευχαριστώ πολύ. Και είμαι και τόσο πολύ έτοιμος που πρέπει να πάω να ψηφίσω σε μισή ε, ώρα για την απόσπαση εργαζομένων και ε, με το ρυθμό που ε, επιβάλλεται ε, ελπίζω να τα καταφέρω και θα τα πω στα ισπανικά. Ευχαριστώ τους και οδησηγητές για τις τροπολογίες και το έργο τους. Πραγματικά βελτιώνουν πολύ το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικά νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε καλούς συμβιβασμούς και το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, έχει και πολλά καλά. Για την αυριανή συνεδρίαση των σκιωδών θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω και να συνενώσω τις τροπολογίες ε, που συμπίπτουν. Βέβαια κάποιες από τις αλλαγές και κάποιες από τις απολογίες θα ψηφιστούν χωριστά. Τι κάνει η πρόταση αυτή, θέτει κοινούς στόχους, ε, υπομορφή αρχών. Άρα, ο στόχος δεν θα πρέπει να ε, θίξει αυτά που ήδη λειτουργούν καλά, αλλά να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε αναδιάρθρωση σωστή, νομική ασφάλεια, δεύτερη ευκαιρία, ασφάλεια δικαίου σε όλη την Ευρώπη και αποτελεσματικές διαδικασίες. Θα ήθελα να σας προτείνω τα εξής. Ε, να τονίσω ε, για το ποιοι είναι οι ενεχόμενοι. Θα πρέπει να ορίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι, εργαζόμενοι και το δημόσιο επίσης θα πρέπει ε, προληπτικά να συμμετέχει στην αδιάρθρωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, αυτοί που συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης θα πρέπει να έχουμε ένα κατάλογο δικτών σε μια ιστοσελίδα για την έγκαιρη προειδοποίηση. Έτσι θα έχουμε περισσότερη ενιαία και εσωτερική αγορά. Δηλαδή θα μοιραζόμαστε τους κοινού ε, στόχους. Το τρίτο, αν θα πρέπει υποχρεωτικά να οριστεί διαχειριστεί ή όχι. Αυτό θα το συζητήσουμε στα διάφορα ε, θέματα που θα δουν οι σκιώδεις ηγητές. Κανονικά το κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει να ε, διορίζεται αυτό για να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των ενεχομένων μερών. Όπως λέει η ίδια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άλλο θέμα, η διάρκεια της ε, αναστολής. Εδώ ε, έχω διάφορες προτάσεις. Είναι της τάξεως μηνών, από τρίμηνο μέχρι εξάμηνο προτείνουν οι διάφοροι σκιώδεις χιτές, αλλά θέλω να μου εξηγήσουν για ποιο λόγο προτείνουν τη συγκεκριμένη διάρκεια ε, στη συνέχεια. Και πιστεύω ότι θα τα βρούμε εκεί. Ε, για την αναστολή και τις ε, συνέπειες, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το γενικό κανόνα που λέει ότι θα ανασταλεί για μια περίοδο η διαδικασία ε, κήρυξη αφαιρεγιότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν δεν ανασταλεί, αν δεν διακοπεί η δυνατότητα να εφαρμοστεί, να επιβληθεί η τότε η ε, οδηγία είναι κενή περιεχομένου και κενή αποτελέσματος. Για ποιο λόγο να προσπαθούμε ε, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να, να το χρέος αν πέσει ο πέλεγης της αφαιρεγγιότητας. Ε, στη συνέχεια, πιστεύουν οι σκιώδεις ότι αρκεί ε, οι βασικές συμβάσεις εκτέλεσης να ε, διατηρηθούν όπως έχουν σε αυτή την περίοδο ή πρέπει να υπάρξει κάποια άλλη ρύθμιση. Τελειώνω. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ε, κατηγορίες και κανόνες για τους εργαζομένους και τους μικρούς παρόχους. Ένα τελευταίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε ε, τι θα γίνει με τα προσωπικά και τα επαγγελματικά δάνεια των επιχειρηματιών, ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως κανόνα, έτσι γενικό, να υπάρχει ενιαία διαδικασία. Αλλά αυτό το βλέπω πάρα πολύ ε, περίπλοκο. και πολύ γενικό. Δεν μπορεί ε, ε, το, το προσωπικό δάνειο να έχει την ίδια μεταχείριση με το επιχειρηματικό. Δεν μπορεί να καταδικάζει τον άλλον και στην προσωπική του περιουσία που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για τους διαχειριστές Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει ε, κάποια προαπαιτούμενα και βασικά κριτήρια ε, γνώση, φήμη, διοντολογία και εκ των υστέρων αξιολόγηση και έλεγχο για τα όσα πράττουν, συλλογή δεδομένων. Επίσης θα πρέπει να σας πω εδώ ότι για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την εφαρμογή της οδηγίας θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσο χρόνο χρειάζεται για την αφαιρεγκαιότητα και την αδιάρθρωση κάθε εταιρεία, να ξέρουμε πόση δουλειά κάνει ο διαχειριστής και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όλα αυτά κατά την άποψή μου σήμερα θα πρέπει να αναγράφονται, να αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Ε, θα βοηθήσουμε λοιπόν όλοι, θα βάλουμε ένα χεράκι να βελτιωθεί το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Τόμ Φαντα Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, υπάρχει εδώ πέρα ένα μεγάλο κοινωνικό στίγμα όσον αφορά την ε, χρεοκοπία περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι στις ε, ΗΠΑ. Θα πρέπει όμως να υπάρξει δυνατότητα με δεύτερες ευκαιρίες. Μία πρόσφατη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου της ε, Γάνδης έδειξε ότι 60% των ατόμων που είχαν χρεοκοπήσει πλέον δεν απολάμβαναν εμπιστοσύνης. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε όσους χρεοκοπούν στις επόμενες ε, πράξεις τους. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ότι οι καλόπιστοι επιχειρηματίες θα έχουν την δυνατότητα με ευκολότερο τρόπο να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, ειδικά για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις ε, και τις μονοπρόσωπες. Πρέπει επίσης να δουλέψουμε περισσότερο στην ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα βοηθάει στην έγκαιρη αναδιάρθρωση αντί για την, ε, το προώρο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Στη Φλάνδρα έχουμε τον οργανισμό που λέγεται Εντίζο που βοηθάει ακριβώς τους ελεύθερους επαγγελματίες ε, σε οτιδήποτε τους ε, δυσκολεύει και κυρίως ε, τους υποστηρίζει στην χρεοκοπία και στην δεύτερη αρχή τους. Ε, και βεβαίως το πρόβλημα εδώ πέρα το μεγάλο είναι ότι συχνά όταν αναγκάζονται οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια είναι πάρα πολύ αργό. Οπότε, όπως λέμε και στο κείμενό μας, σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα να υπάρξει ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης και δεύτερον να υπάρξει σε ένα πρώτο στάδιο, πρώιμο στάδιο, η επαγγελματική συμβουλή των ειδικών. Στις διαπραγματεύσεις τώρα για τις συμβαστικές προτάσεις θα πρέπει να δούμε που, ε, ποιες είναι ακριβώς οι διαφορές στην εθνική νομοθεσία που θα πρέπει να εναρμονιστούν ακριβώς όταν είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για την διάρκεια των διαδικασιών και πρέπει να εναρμονίσουμε εκεί όπου μπορούμε με στόχο να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τους επιχειρηματίες εκείνους οι οποίοι ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να φροντίσουμε να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες εθνικές νομοθεσίες, ε, π.χ. την νομοθεσία περί χρεοκοπίας εάν αυτή λειτουργεί σωστό. Και δεύτερον θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα βρίσκει την ισορροπία μεταξύ πιστωτή και χρεωστή. Γιατί θα πρέπει και οφειλέτη. Θα πρέπει να οδηγηθούμε στην σωστή ε, ισορροπία και βεβαίως ε, αναμένουμε και τις ε, προτάσεις των συναδέλφων για να καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο με βάση την πρότασή του συναδελφού Σαμπον. Σα ευχαριστώ, Τόμ, εξ ονόματο ε, των Σοσιαλδημοκρατών, κυρία Μανταμπέρες. Euh, ε, ζητώ συγγνώμη εξ του συναδέλφου Κοτσολίνο που ε, κολλείται ως Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, εμείς γνωμοδοτούμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες να ασχοληθούμε με τις συνθήκες που επικρατούν κατά την αναδιάρθρωση και να δούμε και την εναρμόνιση του πτωχευτικού δικαίου. Βλέπουμε στα θέματα των τραπεζών πόσο αυτό αποτελεί εμπόδιο. Δεν υπάρχει μια αρμονία ε, στο πτωχευτικό δίκαιο και αυτό είναι ένα βάρος. Ε, κατανοώ όμως ότι όλη η δυσκολία εδώ είναι για το πώς θα προχωρήσουμε αποτελεσματικά. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι χρήσιμη μεν, θα είναι άραγε και ε, ικανοποιητική και επαρκή θα το δείξει αυτό η εμπειρία. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πολύ φιλόδοξο ως προς τους στόχους του. Ε, για τις τροπολογίες λοιπόν που κατέθεσε και ο κύριος Κοτσολίνο αλλά και άλλοι σοσιαλιστές συνάδελφοι να τονίσω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, η διάρκεια. Ένα από τα διακυβεύματα της παρούσης νομοθεσίας είναι ε, να βεβαιωθούμε ότι στα διάφορα κράτη-μέλη οι διαδικασίες πτώχευσης να γίνονται ε, και μετά από συζήτηση, διαφάνεια και αρκετή ειλικρίνεια για να έχουμε και εξαγορές, αλλά και με διαιτησία κάποια στιγμή για να αποφύγουμε να διαιωνίζονται συνεχώς αυτές οι διαδικασίες, ε, ε, πράγμα που κάνει να κινδυνεύουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι προμηθευτές που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των εταιριών αυτών. Επίσης, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες έχουν κάνει τροπολογίες ότι θα πρέπει να μιλάμε ταυτόχρονα και για την αναδιάρθρωση αλλά και για τη μεταβίβαση ε, ταυτόχρονα και ελπίζω και ο εισηγητής να λάβει υπόψη του αυτή την ανησυχία και το μέλημά μας. Τρίτο στοιχείο για τη συλλογή δεδομένων. Βλέπουμε ότι εδώ ε, χρειάζεται οπωσδήποτε κάποια ροή στις πληροφορίες και τα πώς θα γίνει ε, πώς θα βρεθεί μάλλον η ισορροπία ανάμεσα στην ε, ευκρίνεια των διαδικασιών και ε, την επιτάχυνση της μεταβίβασης, γιατί μπορεί στην αρχή να χρειάζεται μία φάση κάπως πιο εχέμηθη, εμπιστευτική, για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες. ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης, μάλλον ε, απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων την περασμένη θητεία, ε, παρακαλώ τον εισηγητή να δει τι είχε κάνει τότε ο συνάδελφος Αλεχάνδρο Θέρκας με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις στην έκθεσή του για το πώς συνδυάζονται αυτές οι διαδικασίες. Διαδικασίες αφαιρεγκαιότητας, εκαθάρισης και συμπερίληψης των εργαζομένων σε αυτή. Θα μπορούσαμε εσείς, τροπολογίες μας, να υιοθετήσουμε μερικά από τα στοιχεία της έκθεσης τέρκα. Ευχαριστώ από την ECR και Τώρα έχεις μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν ΚΕΙ. Ο κύριος Λίντς ε, ζητά συγγνώμη γιατί κολλείεται. Θα διαβάσω την δήλωσή του που δεν περιλαμβάνει ακόμα σχόλια επί των συμβιβαστικών τροπολογιών. Μια γενική σκέψη είναι πολλές από τις τροπολογίες αντικατοπτρίζουν ιδέες που έχουν οι βουλευτές για τα εθνικά καθεστώτα χρεοκοπίας και αναδιάρθρωση. Επίσης, το αρέσει ιδιαίτερα το βελγικό καθεστώς όμως, το θέμα μας στόχος θα πρέπει να είναι να συνδυάσουμε τα καλύτερα στοιχεία σε ένα ενιαίο συνεκτικό σύστημα και το κάθε σύστημα να προσαρμοστεί όπου αυτό είναι αναγκαίο για να γίνει πιο αποτελεσματικό, φτηνότερο και γρηγορότερο. Αυτό πρέπει να γίνει έχοντα κατά νου την πολύ διαφορετική φύση των εθνικών νομικών συστημάτων. Επιπλέον, κάθε τέτοια περίπτωση είναι διαφορετική και για τον λόγο αυτό απαιτείται ευελιξία. Ε, Πηγαίνοντα στι βάθο, ο κ. Λούνε ε, θα ήθελε να πει τα εξή. Πρώτα απ' όλα, μια ενιαία διαδικασία για προσωπικά επαγγελματικά χρέη δεν θα πρέπει να επιβληθεί στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή για εμά. Προτείνουμε να τροποποιήσουμε το άρθρο 23.1 αναλόγως και βεβαίως χαιρόμαστε που υπάρχουν και ανάλογες τροπολογίες. Δεύτερον, ο ορισμός ε, κάποιου ειδικού δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση. Προτείνουμε λοιπόν ε, το πρώτο τμήμα του άρθρου 5 παραγραφής 3 να παραμείνει ως έχει. Δεν είναι πάντα αυτό θετικό ή προς το συμφέρον του οφειλέτη, ειδικά σε περίπτωση που υπάρχουν λίγοι πίστοτες. τρίτων, πρέπει να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για όταν βρεθεί κάποιο σε δύσκολη θέση. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να στέλνουν αυτές τις πληροφορίες στην Κομισιόν για να διευκολύνουν. Με συγχωρείτε. Ο Διερμηνέας είπε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορα, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Τότε να σας παρακαλέσω λίγο πιο σιγά και ξεκινήστε πριν από δύο-τρεις προτάσεις γιατί βεβαίως με ενδιαφέρουν αυτά τα οποία λέτε. Το δεύτερο ή το τρίτο σημείο. Που... Το δεύτερο καλύτερο. Ο ορισμός ε, κάποιου ειδικού δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική. Εδώ πέρα συμφωνούμε με την Κομισιόν και προτείνουμε το πρώτο τμήμα του άρθρου 5, παραγράφος 3, να παραμείνει ως έχει. Μια τέτοια απέτηση βεβαίως δεν είναι πάντα αναγκαία, χρήσιμη ή προς το συμφέρον του φιλέτη, ειδικά σε απλές περιπτώσεις όπου εμπλέκονται λίγοι πιστωτές. Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό για τους επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες εάν βρεθούν σε δύσκολη ή για όταν θελήσουν να ξαναξεκινήσουν. Έχουμε λοιπόν υποβάλει και μια τροπολογία προς τα κράτη-μέλη για να δώσουν αυτές τις πληροφορίες στην Κομισιόν για να διευκολυνθεί η δουλειά της και να μειωθεί το διοικητικό βάρος όταν θα συλλέγουν τις πληροφορίες για όλα τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Λούνες θα ήθελε να πει πως ε, αναμένει να ξεκινήσει η έργαση επί των συμβαστικών τοπολογιών αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και Φαντάζομαι ότι μπορείτε και γραπτό να ανταλλάξετε πληροφορίε παρόλο που θέλετε κάτι στι σημειώσει. Κύριε Βιέγκα, εκ μέρου τη Γκουε. Καλησπέρα. Μόνο μερικέ σημειώσει που μου απεστάλησαν από την συνάδελφο Παλώμα Λόπε. Δύο-τρία λεπτά. Και μόνο βασικά ζητήματα που μα αφορούν στην ομάδα. Πρώτον, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι προτεραιότητα της οδηγίας, δηλαδή να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και οι πιστώσεις τους, που πρέπει να είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων, ισότιμα με τους άλλους, το κόστος και οι απώλειες, η αφαιρεγγιότητα δεν πρέπει να είναι κάτι που θα, τους, θα το υπομειστούν οι ίδιοι. Δηλαδή, στο πλαίσιο οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης, ο ρόλος των εργαζομένων πρέπει να είναι στον πυρήνα, στο κέντρο αυτής της οδηγίας, εφόσον είναι βασικοί πιστωτές. και καθοριστικό μέρος της όλης λειτουργίας της επιχείρησης. Γι' αυτό όλες οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης και αφεντιότητας και απαλλαγής πρέπει να γίνουν σε διάλογο με τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι παρόντες με δικαίωμα βότου, με, με δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα παρουσίας στις συνελεύσεις. Πρέπει επί της ουσίας Αυτά να ληφθούν υπόψη και αυτά ήθελε η συνάδελφο Παλώμα Λόπε να ακουστούν εδώ. Ότι οι εργαζόμενοι είναι ε, αναπόσπαστο τμήμα μια επιχείρηση, οι πιστώσει του πρέπει να ε, προστατεύονται με τη δική του τη φωνή που θα πρέπει να ακούγεται σε κάθε διαδικασία αναδιάρθρωση και πρέπει να παραμείνουν στο κέντρο των μεριμνών αυτής της νομοθετικής πρότασης γενικώ. Ευχαριστούμε. Από τους Πρασίνους θα μιλήσετε εσείς εκ μέρους του κύριου Γκίγκολντ. Ναι, θα σας διαβάσω την εξή δήλωση. Καλωσορίζουμε τη βασική, το βασικό στόχο της οδηγίας αυτής να άρει τους βασικούς φραγμούς στη διασυνοριακή ροή κεφαλαίων από τα διαφορετικά πλαίσια αναδιάρθρωσης των κρατών μελών. Θέλουμε να δημιουργηθεί μια διαδικασία ελάχιστων προτύπων, ε, νομικώς δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη. Στι ε, διαδικασίε αναδιάθρωση και φερεγγιότητα πρέπει να υπάρξει καλή εξακολούθηση τη λειτουργία μια επιχείρηση, οπότε να μην ε, σωρευθούν δάνεια τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, που πιέζουν τον τραπεζικό κλάδο. Αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά του και τι προσπάθειέ του να συμπληρώσει την πρόταση τη Επιτροπή. Επίση, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι κάποιε από τι τροπολογίε μα έχουν συμπεριληφθεί στι συμβαστικέ λύσει που κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα, ιδίω ό,τι αφορά πρώτον την ενίσχυση του συστήματο έγκαιρη προειδοποίηση και των σχετικών δικτών που μπορούν να σημάνουν αρνητικέ εξέλιξει στη λειτουργία μια επιχείρηση και δεύτερον τη συλλογή ε, δεδομένων και το σύστημά τη. Βεβαίω, υπάρχει ένα φάσμα ζητημάτων που είναι σημαντικά και δεν έχουν αντιμετωπιστεί και θα, πρέπει, να, θα πρέπει να τα προσέξουμε. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στι προσπάθειέ μα, να προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στι διαδικασίε αναδιάρθρωση ε, και και έγκαιρης και θα πρέπει να προβλεφθούν και κατάλληλε διαδικασίε. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε αποτελεσματικά το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση, διαβούλευση και συμφωνία σε όλε τι φάσει τη διαδικασία. Σημαντικό είναι οι εργαζόμενοι χωρίς όρου να εξαιρούνται οποιαδήποτε διαδικασία αναδιάσωσης. Δηλαδή να μην είναι η επίδοση της εταιρεία όρος για την σύναψη του συμβολέου τους και να μην χάνουν τα χρηματικά τους δικαιώματα και να μην υπάρχει παρέμβαση στο θεμελιώδε δικαιώματα τη ε, ελευθερία στην απασχόληση. Επίση, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα ελάχιστη εναρμόνιση, όπω προτείνει η οδηγία, αλλά δυστυχώ η προσέγγιση δεν είναι σφαιρική στο να εναρμονιστούν νόμοι αφαιρεγκαιότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι βασικέ πτυχέ του νόμου περί αφαιρεγκαιότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα τη ρήτρα ε, αναθεώρηση και να συμπεριληφθεί στην οδηγία. Πρέπει όλες οι επακτικές και νομικές προκλήσεις που μας απασχολούν να αντιμετωπιστούν με την ίδια ε, σφαιρική προσέγγιση και να υπάρχει φιλοδοξότερη δράση ώστε να ορίσουμε κοινό έδαφος για την αναδαμόνιση των νόμων των κρατών μελών για την αφαιρεγκαιότητα. Πρέπει να υπάρχει συνολικότερα εναρμόνιση ώστε να ε, λειτουργήσει πιο ε, αποτελεσματικά και εύρυθμα και η αγορά κεφαλαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Και τελευταίο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Θέλετε να πείτε λίγα λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα να, αντιμετωπίσω, να απαντήσω στα θετικά σχόλια και σε κάποιες από τις ανησυχίες για την πρόταση. Ε, χαίρομαι που υποβάλλατε τις προτάσεις σας για το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης. Είμαστε ανοιχτοί στο να αποσαφηνίσουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό, ο λόγος που δεν το κάναμε είναι επειδή σε μερικά κατημέλη δεν έχουμε στοιχεία για το σύστημά του. Θέλαμε λοιπόν να παραμένουμε ευέλικτοι. Ω προ τη συλλογή των δεδομένων, καλωσορίζουμε τη θετική αποδοχή τη πρότασή μα και βεβαίω θα πρέπει να δούμε και το κατά πόσον χρειάζονται ή όχι ειδικοί στα θέματα αυτά. Εάν πρόκειται για μια μικρομεσαία επιχείρηση, σίγουρα θα πρέπει να παρέμβει ένα ειδικό, γιατί η, η μικρομεσαία αποκλείται από τη διαδικασία αναδιάρθρωση. Και μετά για την ενιαία διαφορετική μεταχείριση των καταναλωτών και επαγγελματικών δανειών, των καταναλωτικών επαγγελματικών δανειών. Όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση καταναλωτικών και επαγγελματικών δανείων. Ε, μάλλον στα επαγγελματικά τίνει να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση. Γι' αυτό παραμείναμε στα επαγγελματικά δάνεια, γιατί μπορούμε να ρυθμίσουμε το κόστος της όλης διαδικασίας. Και η παρατήρηση για την προστασία των εργαζομένων, η πρόταση οδηγίας που κάναμε, προβλέπει την συμμετοχή των εργαζομένων στις διαβουλεύσεις και η προστασία τους είναι σαφή. Δεν θέλαμε να αλλάξουμε κανένα από τα δικαιώματα που ήδη έχουν βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Οπότε εδώ το θέμα αυτό διευθετείται πιστεύω. Οι εργαζόμενοι διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους βάσει των όσων ήδη ισχύουν και σε σύγκριση με αυτό το νέο μηχανισμό αναδιάρθρωσης. Και τέλος, για την ευελιξία και την γενική δομή του συστήματος. Είναι πολύ δύσκολο. Να πάρουμε τα καλύτερα των καλύτερων από τα παραδείγματα, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν κάποιε ελάχιστε απαιτήσει με αρκετό περιθώριο για τα κράτη-μέλη να κινηθούν εντό των ορίων που έχουμε προδιαγράψει είναι μια συμβαστική λύση μεταξύ της απόλυτης ε, διαλλακτικότητας και του να έχουμε ελάχιστα πρότυπα, κοινά πρότυπα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα συνδυάσουμε όλα σε συστημικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν δύο ολόιδια συστήματα αναδιάρθρωσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κάτι μέλη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και να ρωτήσουμε και τον εισηγητή αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, θέλω Βεβαίως. Αύριο έχουμε τη συνεδρία των σκιωδών, θα κάνουμε καλή δουλειά και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο γιατί όλα αυτά που άκουσα είναι επικοδομητικά, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Συμφωνώ με το φίλο Τόμ Βαντεκέντελάρα. Η ουσία ίδια είναι ακριβώς αυτή, να σώσουμε την εταιρεία, τον επιχειρηματία και κυρίως να μην τον στραγγαλίσουμε ε, και την επιχείρησή του. Αυτό θα κάνουμε. Συμφωνώ επίσης με την κυρία Μπερές και εκεί που μίλησε για διαφάνεια, για να αποφύγουμε ε, διαδικασίες χωρίς ισορροπία, να λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες διαδικασίες, δεδομένα, όλα αυτά. 30 χρόνια φιλίας με συνδέουν με τον Αλεχάνδρο Θέρκας. Πολύ ε, κοντά ε, είναι το γραφείο του στο δικό μου γραφείο και το σπίτι του και θα συναντηθώ μαζί του πριν ε, συνεδριάσουμε με τους σκιώδεις συγητές. Και πραγματικά θα υιοθετήσουμε πολλά από τη ενδιαφέροντα της έκθεσης. Το ECR μα δίνει και καλέ ιδέες σε τεχνικό επίπεδο. Θα πρέπει να το κοιτάξω αυτό το 23 που λέτε. Έχουμε ε, πολύ καλή τεχνική συνεργασία, επαναλαμβάνω, αλλά πάντα το πρόβλημα ποιο είναι. Εμείς είμαστε πιο κοντά στην περισσότερη Ευρώπη από ότι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Αυτό είναι ε, χαρακτηριστικό μας. Ε, Κατανοώ τα όσα λέει ο κύριος ε, Βιέγκας και ευχαριστώ και τον κύριο Ορτάσον για τα καλά του λόγια. Και όπως η κυρία Μπερές και ο κύριος Βιέγκας επέμεινε ε, στο πρόβλημα, που δεν είναι ακριβώς το πρόβλημα, στο ρόλο θα έλεγα των εργαζομένων. Βεβαίως θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Βεβαίως και εγώ είμαι υπέρ της περισσότερης Ευρώπης όταν μιλάτε για μεγαλύτερη εναρμόνιση. Ενδεχομένως εμείς να το προτείνουμε, αλλά όχι στο βαθμό που να σπάσουμε το συμβιβασμό και την ισορροπία σε μια τεχνική θέση λόγω αυτού. Δεν θέλω να διχαστούμε. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν περισσότερο από μένα στην επικουρικότητα. Μια που μιλούμε για τους εργαζομένους, να πω τα εξής δύο. Πρώτον, η απασχόληση και ο Γιώργη Μουσκιώδης ενέκρινε αυτά τα στοιχεία, Επιτροπή Απασχόλησης δηλαδή. Ε, μπορούμε να ε, ε, υιοθετήσουμε κάποια από τα όσα μας έχουν προτείνει και εκείνοι. Και ένα δεύτερο, θέλω να σας θυμίσω ότι εδώ μιλάμε κυρίως για την οικονομική, χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και υπάρχουν ειδικοί νόμοι για την κατάσταση των εργαζομένων, για την κατάσταση των πιστωτών ε, στην Ισπανία ας πούμε υπάρχουν ε, ειδικέ ρυθμίσεις και, είναι συγκεκριμένοι οι φορείς και ε, οι πιστωτές και οι οφειλέτες. Συμφωνώ με όλα αυτά που λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή των εργαζομένων κτλ. Δεν έχει νόημα να αποστούμε έστω και ένα χιλιοστό από τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα το καταπολεμήσω και θα αγωνιστώ εγώ εκεί για την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ και την Κομισιόν και τους Σκιώδης και όλους τους συναδέλφους. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είμαστε ακριβώς στις 5 ε, και 4, όπως ζητήσατε. Ε, τηρούμε το χρόνο διαγράμμα μας. 6 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, 7 Νοεμβρίου στη Γιούρη λίγη προθεσμία 20 και 21 Νοεμβρίου θα το εξετάσει η Επιτροπή Γιούρη και η ψηφοφορία θα γίνει το Ιανουάριο. Διάλειμμα και πάλι 25 λεπτά πριν τις ψηφοφορίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε τις ψηφοφορίες μας με την κλασική δοκιμή. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα δοκιμαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. You abstain. I always abstain at test. Ο Μπράνα που έχει θα ψηφίσει σχεδόν πάντα, λέει ο κ. Φέρβερ. Press the button, Brian. Bravo. yes, sir, I'm hoping this is Okay. Close. Ένας λοιπόν της ψηφοφορίας. Καλώς. Αρχίζουμε λοιπόν. Έκθεση του κυρίου Χοκ, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, Οικονομικέ πολιτικέ τη ζώνη του ευρώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, παρακαλώ, πριν μπούμε στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε μια πολύ ε, καλή και πολύ ωραία συνεργασία για να φτάσουμε στους ε, συμβιβασμούς. Ευχαριστώ όλους και όλους τους για τις προσπάθειές τους. Το εκτιμώ βαθύτατα και πραγματικά κάτι καταφέρνουμε όλοι μαζί από κοινού. Το πρόβλημα είναι η διαδικασία γενικότερα, έτσι, ευρύτερα. Εκτός από την έκθεση αυτή, έρχεται να προσθεθεί και μία άλλη από την Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία ανακοινεί άλλα ζητήματα που δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τις συστάσεις αναχώρα και τη συνέχεια που δίνεται στην οικονομική πολιτική. Και αυτό μας προβληματίζει. Δεν χρειάζεται να το δούμε σήμερα. Θα πρότεινα να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Απλώς θέλω να σας ανακοινώσω ότι τώρα έχουμε ειδικέ ανάγκες δημιουργήσει για την Ολομέλεια. Αυτό που θα ήταν πολύ άνετο και απρόσκοπτο Τώρα δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί έχουμε δύο εκθέσεις, μία που δεν έχει ζητηθεί καθόλου, δεν έχει τύχει διαπραγμάτευσης, δεν έχει μπει στη διαδικασία, δεν το έχω δει ούτε εγώ τη Σκιώδης το κείμενο ότι η Επιτροπή μας και επηρεάζει όμως από την άλλη ε, πολιτικές ε, και δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με την οικονομική πολιτική της συστάσης αναχώρα και τι να κάνουμε θα πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα στο μέλλον γιατί δεν είναι διαδικασίες αυτές που μπορούμε να επιτρέψουμε και να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ασημερίζομαι τις ανησυχίες σας. Για το λόγο αυτό επιμένουμε ακριβώς για να βελτιώσουμε τη δομή για την έκθεση αυτή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το σημερινό σύστημα που κινδυνεύει να οδηγήσει σε κάποιες αναντιστοιχίες όταν δύο, πράγμα, δύο επιτροπές συζητούν το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι συμφωνούμε και θέλουμε και οι δύο να βελτιώσουμε την κατάσταση για το μέλλον. Για την Ολομέλεια οι πολιτικές ομάδες είναι κυρίαρχες ότι θα αποφασίσουν πολιτικά αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ας ε, ψηφίσουμε συμβαστική τροπολογία α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 73 ψηφί περ κατά έλεγχος παρακαλώ για την τροπολογία 73. Ψηφίζουμε. Περάσει τη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική E υπέρ ε κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 216 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Η 220 υπέρ κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Αν θέλετε να το ελέγξουμε, το ελέγχουμε, αλλά μου φαίνεται είναι σαφέ. Συμβαστική. Εν. Ποιο ζητάει έλεγχο, ζητά έλεγχο, όχι. Εν υπέρ, κατά, άποχέ, ε, εγκρίνεται. Συμβαστική ο, μικρόν υπέρ, κατά, άποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 345 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε, Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται η τροπολογία 407 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα αυτό τώρα τι είναι εδώ. Εδώ έχει ένα θετικό πρόσημο, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Okay. Do not λοιπόν, δεν ψηφίζουμε τις Επιτροπής Απασχόλησης και θα ψηφίσουμε μόνο Ρέτζι 1, τροπολογία 1 της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι στη σελίδα 36, λέει ο πρόεδρος του δικού μου καταλόγου. Μετά τα έμπλ λέει κάπου Ρέτζι. Τροπολογία 1 είπε, κατά έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Vote is closed. Απορρίπτεται. Ρέγγι 2. Μόνο το τελευταίο τμήμα. Τελευταία πρόταση υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι στην παράγραφο 8 υπέρ κατά έλεγχος. Αρχίζει τώρα για την πρόταση της Επιτροπής Ρέζη στην παράγραφο 8. Απορρίπτεται. Ρέτζι 9 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι παράγραφος 12 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 14 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ονομαστική κλίση τώρα για το σύνολο του κειμένου που τροποποιήθηκε. Αρχίζουμε τώρα. Πέρας. 33 υπέρ, 8 κατά και 5 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε εισηγητά μου. Και στην ομάδα διαπραγμάτευσης αξίζουν. Συγχαρητήρια. Τώρα έχουμε μια σειρά έγκαιρων ε, μη ε, ε, αντιρρήσεων που έχουν συμφωνήσει ε, οι εισηγητές και οι συντονιστές της Επιτροπής μας και έχουν νόημα πιστεύουν. Α, εγώ ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή όμω, γιατί θα ψηφίσουμε τη δική σας έκθεση. Κύριε να έχετε το λόγο. Σύντομα θέλω να πω κάτι για τις δύο προτάσεις για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Κανονικά επί της ουσίας είναι εντάξει και οι δύο, αλλά ήδη ε, από το Μάιο-Ιούνιο και μετά Ιούνιο-Ιούλιο και τελικά στις 21 Σεπτεμβρίου έφτασαν οι προτάσεις. Προτείναμε ο Πρόεδρος και εγώ να παρακαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να έρθει με διαφορετική νομοθετική πρόταση για να μεταθέσει την 1η Οκτωβρίου 2018 να παρατείνει την προθεσμία για τους χρήστες. Ε, όχι για τα κράτη-μέλη, 23 ε, να Φεβρουαρίου συγγνώμη, να παραμείνει, αλλά για τους πελάτες, ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους, να παραταθεί η προθεσμία. 1η Οκτωβρίου 2018 και παρακαλούμε να συμφωνήσετε γιατί ορισμένα κράτη-μέλη μας δηλώνουν ρητά ότι δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά και έχει τα κράτη εταιρείε βασικά. Ευχαριστώ πολύ. Μερές. Η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα υποστηρίξει την πρόταση του εισηγητού. Να σας πω για ποιο λόγο φτάσαμε ως εδώ, γιατί ζητάμε αυτή την παράταση. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε κατεξοδότηση πράξης ε, ζητούμε να υπάρξει ένα διάστημα από την αρχή ε, Τη θέση σε ισχύ της κατεξουδότηση πράξης μέχρι την νομοθεσία, ένα εξάμεινο. Αλλά τώρα έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε μας αναγκάζει να ζητήσουμε αναβολή της θέσης σε ισχύ ε, της ίδιας της νομοθεσίας. Αυτό είναι λυπηρό ως κατάσταση και φυστούμε την προσοχή στους ηθήνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε στο μέλλον να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο γιατί κάθε φορά το Κοινοβούλιο θα ζητάει αναβολή ε, τη ισχύω τη νομοθεσία. Αν δεν προβλέπετε το εξάμεινο, Εκτό αν είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ε, δεν προϊονίζεται τίποτα το θετικό για το μέλλον. Σαφέ λέει ο κύριο Λάνη. Σε ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον να αναστάει το λόγο, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτα, όλα πρέπει να ψηφίσουμε ένα την παράγραφο Τώρα μιλάμε για την μη υποβολή αντίρρησης ε, στο IDD για τις ε, διατάξεις που αφορούν τις ασφαλιστικές εταιρείες ανεξαρτήτως ε, σύμφωνα με τον κανονισμό της 21 Σεπτεμβρίου 2017 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τις ιδεολογικές γεύσεις υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 επί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. 41 υπέρ 3 κατά 2 αποχές. Περνάμε στην δεύτερη πράξη εξουδότηση. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, αρχικό κείμενο παράγραφος 1-2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές αν μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εκτιμώντας α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ 4 κατά δύο αποχές συγχαρητήρια και νομίζω ένα σαφές μήνυμα για λόγους βεβαίως που μας ε, λυπούν και θα πρέπει να αποφευθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, δεν είναι η πρώτη περίπτωση. Είχαμε αναβολή και ίσως και μεγαλύτερη αναβολή από αυτήν. Οπότε αφενός πρέπει να αποφευχθεί η επανάληψη αυτού του πράγματος. Από την άλλη ελπίζω η Κομισιόν να ακολουθήσει την Συμβουλή του Κοινοβουλίου και την αξιολόγηση του εισηγητή για την αναβολή αυτή που είναι αιτιολογημένη. Και ούτως ή άλλως τώρα έχει και τη στήριξη της Επιτροπής. Τώρα ψηφίζουμε την διαδικασία μια για έναν ε, κανονισμό της Μίφιντ Μάρκους. Έχετε τον λόγο να ευχαριστώ. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω πως ε, υπήρχε μια τεχνική συμβουλή που έδωσε η ΕΣΜΑ στην Κομισιόν πριν από ένα έτος ε, και παρέμεινε εντός Κομισιόν και εκτός κάποιων συντακτικών αλλαγών δεν έκανε τίποτα η Κομισιόν και τώρα ζητάμε να κάνουμε αυτή την κίνηση γιατί είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν τα συστήματα και είναι απαράδεκτο να περνάει ένας χρόνος χωρίς ε, καμία ουσιαστική αλλαγή στην τεχνική συμβουλή της ΕΣΜΑ. Η Κομισιόν έπρεπε να το έχει κάνει πολύ νωρίτερα και δεν θα είχαμε τώρα αυτή την χρονική πίεση. Αυτά μόνο για να είστε ενημερωμένοι. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Ναι. Λογικό φαίνεται. Οπότε, σφίσμα μπλοκ της παραγράφους 1 και 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογικές αναφορές υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εκτιμώντας α υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εκτιμώντας β υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εκτιμώντας γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται εκτιμώντας δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Το κείμενο στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 41 υπέρ 4. Κατά μια αποχή εγκρίνεται τώρα. Τέλος. Ναι περνάμε σε άλλη μία παρόμοια διαδικασία και αφορά την έμεση εκαθάριση. Δεν ξέρω αν ο κύριος Λάγκεν έχει κάποιες παρατηρήσεις να κάνει. Είναι το ίδιο θέμα που είπε ο κύριος Φέρμπερ, το ίδιο πρόβλημα. Έπρεπε να έχει συμβεί πολύ νωρίτερα. Έχουμε τώρα το Refit και έρχεται μία πράξη Κάτι εξουσιοδότηση. Πρέπει να πιέσουμε να έχουμε μια καλύτερη διοργανική συμφωνία με την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ναι, σαφώς έχει παρατραβήξει. Λοιπόν, παραγραφή 1 και 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται αιτιολογικες αναφορέ. αναφορές 1-9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνονται εκτιμώντα α υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται νομίζω μπορούμε να τα ψήσουμε και τα εκτιμώντα υπέρ ε, κατά αποχέ εγκρίνονται το κείμενο σύνολό του άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία και πέρασε 41 υπέρ 4 κατά μία αποχή εγκρίνεται συγχαρητήρια. Τελείωσαν οι οι και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ποιος θα προεδρεύσει εγώ φοβάμαι. I Fine. Okay, so now we are. Uh, yes, uh, we move to point 13 of the agenda. Περνάμε στο σημείο 13 της σημερινής διάταξης. Καταπολέμηση νομιμοποίησης εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Όπως γνωρίζετε αυτή είναι μια γνωμοδότηση καθότι η αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕΡ, Η κυρία Βαζολή είναι, είναι συντάκτρια μάλλον, της 69 ετροπολογίες Θα της δώσω μέσα το λόγο. Yeah. Παρακαλώ κυρία Βαζολή, έχετε το λόγο. Για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, με τους οποίους συνεργαστήκαμε για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Ήταν πολύ γόνιμη η συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο, στη περασμένη Ολομέλεια και νομίζω ότι και οι συμβιβασμοί είναι εξαιρετικοί. Εκτός από τις συμβαστικές τροπολογίες που σας προτείνω, θα ήθελα να τονίσω μερικά σημεία ε, τα οποία ε, κατά την άποψή μου θα πρέπει να προσθεθούν στη γνωμοδότησή μας. Το φορολογικό έγκλημα ε, είναι, είναι βασικό και θα πρέπει να τιμωρείται με τουλάχιστον φυλάκιση ενός έτους. Ορισμένα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν προβλέψει στην νομοθεσία τους τη φυλάκιση για ε, φορολογικά εγκλήματα. Αλλά ε, ανεξαρτήτως των κυρώσεων θα πρέπει να θεωρείται βασικό. Στην παράγραφο κεφάλαιο 5 παράγραφο 2 προτείνω η φυλάκιση ε, μέγιστη να είναι όχι τετραετής αλλά πενταετής γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα δικήματα. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε και ένα ανώτατο όριο ε, για αυτοργία ε, με διάφορους τρόπους που θα πρέπει να, να αυτοργία να είναι μέχρι τριετία. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν χαμηλότερες ποινές για την ε, προώθηση, υποβοήθηση και ε, ηθική αυτοργία, αλλά βεβαίως αυτό είναι απόκειται στα κράτη-μέλη, ε, αν θέλουν να τιμωρείται λιγότερο ο ηθικός αυτοργός από το φυσικό. Τώρα, για τις υπόλοιπες κυρώσεις. Mm. Απαγόρευση εισόδου ε, ε, συμμετοχής μάλλον σε διαγωνισμούς για δημόσιες προμήθειες ή αποκλισμός από ε, την επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τις, τα, τις καταστάσεις που επιβαρύνουν την υπόθεση, είναι η τρομοκρατία Εκεί επίσης όταν ε, ε, πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο, ένα, δημόσιο που έχει, ένα πρόσωπο που έχει έκθεση σε δημόσια καθήκοντα. Ε, έχει, εδώ έχει να κάνει με ένα θέμα επίσης με τις εξουσίες που έχουν τα κράτη-μέλη να προχωρούν σε άσκηση δίωξης. Υπάρχει μια ανασφάλεια ε, δικαίου θα πρέπει να βάλουμε μια ταξινόμηση προτεραιοτήτων στους διάφορους ε, τομείς που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Πρώτον, η επικράτεια στην οποία έχει διαπραχθεί ε, η αξιόπινη πράξη. Δεύτερον, η εθνικότητα του δράστη. Τρίτον, η χώρα προέρευσης και τέταρτον, η χώρα σύλληψης του ή εντοπισμού του. Επίσης προτείνω να προσθεθεί Ε, να προσθεθεί η δυνατότητα να προσφεύγουμε στη Eurojust για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ε, προσβλέπω στην υποστήριξή σας ε, για τις συμβιβαστικέ προτάσεις και περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσω τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Τόμας Μάνεβε. Υπάρχει κάποιος από το ΕΛΚ ε, που θα εκπροσωπήσει τον κύριο Μάν. Όχι. Για τους σοσιαλδημοκράτες λοιπόν, Υγμπαγέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι ένα άκρο σημαντικό θέμα. Ξέρουμε τα προβλήματα που δημιουργεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ξέρουμε πώς μπορεί το οργανωμένο έγκλημα να ε, ξεπλένει αστρονομικά ποσά. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η πρόταση αυτή οδηγία για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματο είναι ήδη ένα το βήμα, αλλά δεν έχουμε καλύψει όλα τα θέματα. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόταση της Επιτροπής που ευνοεί την διακρατική συνεργασία με ελάχιστου κανόνε ό,τι αφορά τον αντοπισμό των αδικημάτων και τι ενδεχόμενε ποινικέ κυρώσει στον τομέα του ξεπλήματο. Το, το κείμενο αυτό τη Επιτροπή είναι μια καλή βάση εργασία και οι προτάσει τροπολογιών της συναδέλφου Ζολή, ενισχύουν τα θεμελή του κειμένου. Εφόσον θα διευρύνουμε τον ορισμό των αφορολογικών αδικημάτων που συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητε του οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό το ξέπλυμα, με 3 6 χρόνια κάθριξη για, τη, για τους όλα αυτά ε, τα καλωσορίζουμε καθώς δεν θα είναι τα αποδεικτικά στοιχεία απαραίτητο εμφανή ε, εφόσον υπάρχει εικασία για ε, δραστηριότητα ξεπλήματος και επίσης θα υπάρχει διακριτή αντιμετώπιση με μέγιστη ποινή για τις ε, διαδικασίες του, της απάτης και τον απότερο σκοπό του ξεπλήματος και μετά η διαφορά φυσικού και νομικού προσώπου την επιβολή ποινών. Πάντω, πρώτα δεν θα μακρηγορήσω γιατί έχουμε πολύ θετική αποτίμηση για το όλο θέμα. Στην τελευταία συνάντηση των σκιωδών και το κλίμα ήταν πολύ θετικό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λού και ε, εκ μέρου του κύριου Φόξ. Ευχαριστώ και εκ μέρου του κυρίου Φόξ να διαβάσω και εγώ το σημείωμά του. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Υπέβαλα τροπολογίες με σκοπό να έχουμε μια αναλογική προσέγγιση και τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν ε, μέτρα σε εθνικό επίπεδο εφόσον τα επιθυμούν. Οι άλλες ομάδες έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζουν τις τροπολογίες με αφορμή τις εκθέσεις για την Πάνα και θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει την, ε, τις FAF αλλά εμεί θα λέγαμε να μην διαπρέμε τόσο πολύ το πεδίο τη συγκεκριμένη πρόταση. Υπάρχουν πολλέ τροπολογίε που η δική μα ομάδα δεν μπορεί να δεχτεί. Τα φορολογικά παραμένουν αρμοδότητα των μελών και δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το κείμενο. Το να μειωθεί το όριο των μετόχων από το 25% δεν είναι εφικτό, ούτε χρειάζεται η οριζόντια προστασία των ε, καταδοτών σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται μια ε, ισόρροπη προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρξουν ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η ομάδα μου ε, είναι γενικώ επιφυλακτική για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Θα το συζητήσω με συναδέλφου και θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε τροπολογίε. Ανυπομονώ για τη συνεργασία με του τι επόμενε εβδομάδε. Αυτά ω προ τι δηλώσει του κυρίου Φόξ. Ε, Προσωπικώ να προσθέσω ότι ότι σε ένα σημείο ως προς την άποψη του κυρίου Φόξ ε, για τη μείωση του επίπεδου του, του, ορίου των μετόχων από 25% θεωρώ ότι είναι όχι μόνο εφικτό αλλά και επιθυμητό. Και επίσης η προστασία των καταγγελόντων είναι σημαντική υποχρέωση του Κοινοβουλίου. Οπότε σε αυτά διαφωνούμε με τον κύριο Φόξ. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση ότι όλα αυτά δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. και δεν μπορεί να υπάρχει οικονομικό όφελο από την αποκάλυψη πληροφοριών από την πλευρά των καταγγελόντων. Πάντως κάτι πρέπει να κάνουμε για την προστασία αυτών των ανθρώπων ούτω ή άλλω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επειδή συζητάμε για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και για τους καταγγέλλοντες. Μάθαμε η Δάφνη Καρουάνα από την Γαλίτσια, Μάλτα. από τη Μάλτα, έχασε τη ζωή της από βομβιστική επίθεση στη Μάλτα. Θλιβερέ ειδήσει. Συμμετείχε στι όλε έρευνε για την Επιτροπή Πάνα. Την είχαμε ακούσει. Ε, εκφράζουμε λοιπόν την έντονη καταδίκη μας για αυτό το γεγονός. Για την άλλη δεν βλέπω κανέναν. Α, η Βαζουλή. Ναι, τι, να σας δώσω το λόγο, ναι. Μπερδεύτηκα. Ε, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουμε τους κέντρους εισηγητές. να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Γερόν Μπλούσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα είναι θλιβερή η είδηση και τα δικά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της ε, δημοσιογράφου και βεβαίως και η προστασία των πληροφοριοδοτών είναι κάτι που απασχολεί την Κομισιόν, αλλά πρέπει να το δούμε με τρόπο οριζόντιο και όχι μόνο στο πλαίσιο του οικονομικού εγκλήματος. Επίσης, ε, να αναφερθώ σε κάποια σχόλια που γίνονται ότι η οδηγία αυτή συμπληρώνει το προληπτικό πλαίσιο που επανεξετάζουμε αυτή τη στιγμή σε τριμερείς διαλόγους. Θεωρούμε ότι κάποιες από τις τροπολογίες καλύτερα θα ε, τέριαζαν εκεί. Οπότε πρόκειται για μια απάντηση στο ξέπλυμα χρήματος. Ορίζει το αδίκημα και τις σχετικές ε, κυρώσεις. Εκτιμούμε την στήριξη για τα βασικά στοιχεία της πρότασης και βεβαίως το πεδίο εφαρμογή θα πρέπει να διευρυνθεί για να περιλάβει όλα τα σοβαρά δικήματα. Όπως είπε η κυρία Ζολή, η πρότασή μας περιλαμβάνει και φορολογικά δικήματα και είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε πώς μπορεί να έχει έναν πιο έντονο ρόλο στην οδηγία. Η πρώτη αξιολόγηση είναι θετική, παραδείγματο χάρη, ε, με το να διευρύνουμε τις ποινές έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και την φυλάκιση για να υπάρχει αποτρεπτικός χαρακτήρας. Επίσης, ε, με το να μειώνουμε τα εμπόδια όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές υποθέσεις και ελπίζω βεβαίως να ξεκινήσουν προσεχώς και οι διοργανικές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα η κυρία Ζολή για τις τελευταίες της παρατήρησεις. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τα σχόλιά σας. Νομίζω θα διοργανώσουμε την άλλη εβδομάδα μια τελευταία συνεδρίαση των σχεδόν στο Στρασβούργο όπου μπορούμε να ακούσουμε τις διάφορες ε, προτάσεις και γνώμες. Την περασμένη φορά ήταν ευρύτατη η συμφωνία και η συναντήληψη. Και πραγματικά τα φορολογικά εγκλήματα θα πρέπει να θεωρούνται βασικά κύρια εγκλήματα. Ήταν ε, τεράστια το κενό αυτό που υπήρχε στην νομοθεσία. Ε, βεβαίως ε, το ξέπλυμα χρήματος είναι εξώπινη πράξη, αλλά δεν ήταν κύριο έγκλημα. Και στην οδηγία για την καταπολέμηση νομιμοποίησης ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι φρικτό αυτό που μάθαμε για το θάνατο της δημοσιογράφου από τη Μάλτα, την οποία συναντήσαμε στην αποστολή μας στη Μάλτα, την αποστολή ε, την ερευνητική, εξεταστική των πραγμάτων, δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση του ξεπλήματος ε, του χρήματος και θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον κοινέ ελάχιστες κυρώσεις για να αυξήσουμε την πίεση και να ανεβάσουμε τον πύχη. Είναι ακριβώς το κέντρο των παρανόμων ε, ροών κεφαλαίων που προέρχονται από κάθε είδου εγκληματικέ δραστηριότητε, ακόμα και τρομοκράτε ε, χρηματοδοτούνται έτσι. Έχει έρθει η στιγμή να νομοθετήσουμε και μάλιστα αυτή η νομοθεσία να είναι δεσμευτική και πάρα πολύ καλή. Ε, προσβλέπω λοιπόν στην επόμενη συνεδρίασή μα και την περιμένω με χαρά. Ευχαριστώ. προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Μάλλον, στις 6 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, στις 20 Νοεμβρίου. Έτσι, μπορούμε τώρα εδώ να κηρύξουμε το πέρα στη συνεδρίασή μας, αφού σας πω ότι η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα την 5η 19 Οκτωβρίου, 9 με 12.30 το πρωί. Ευχαριστώ.